Colleagues, let us start. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε τρεις ακροάσεις σήμερα στο πρόγραμμα. Το πρώτο σημείο μας σε διάταξη αφορά την έγκρισή της. Υπάρχουν μήπως σχόλια για το σημείο αυτό. Για την έγκριση δηλαδή της ημερήσιας διάταξης. Όχι. Οπότε εγκρίνεται. Όπως πάντα η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο και διερμηνία έχουμε ε, σε 20 γλώσσες. Η αποφάση των συντονιστών της 22ης Ιανουαρίου του 2020 θα αποστελούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ε, απεστάλησαν μάλλον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη σε 6 Φεβρουαρίου. Και πάμε κατευθείαν στο σημείο 3 που αφορά την παρουσίαση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών των δύο εκθέσεων για το blockchain και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζουμε να μάθουμε πολλά από τις ε, παρουσιάσεις σας. Ε, καλωσορίζω τον κύριο Αλεξάνδρ Πολβορά και τον κύριο Μάσιμο Κράλια από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Υπηρεσία Γνώσης και Επιστήμης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που προσφέρει ανεξάρτητες επιστημονικές γνωματεύσεις και υποστήριξη στην ευρωπαϊκή πολιτική. 45 λεπτά, 3 τέταρτα προβλέπονται για την εξέταση των δύο αυτών εκθέσεων του Κοινοκέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακαλώ οι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν μέρος μετά στη συζήτηση να μας το δηλώσουν για να σας σημειώσουμε. Σηκώστε κάθετα την ταμπέλα του ονόματό σα για να σημειώσουμε στο κατάλογο των ομιλητών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στου κυρίου Πολβορά και Κράλια για τι παρουσιάσει σα. Έχετε από 6 λεπτά ο καθένα και θα ακολουθήσει γύρω με του συντονιστέ που θα μιλήσουν για 2 λεπτά ο καθένα. Α ακούσουμε όμω πρώτα τι ομιλίε των εμπειρογνωμόνων μα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την πρόσκληση. Ε, ήταν, είναι περσινή η έκθεσή μας για το blockchain. Η πρώτη παρουσίαση έγινε τον Σεπτέμβριο και μάλιστα έξι τμήματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών συνεργάστηκαν και με τις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ εντοπίζουμε πολλές ε, επαναστατικές αλλαγές και επίσης χρησιμοποιούμε μια συμμετοχική προσέγγιση και αναλύουμε τις διάφορες τάσεις. Καταρχήν, ένα ε, σύντομο σεμινάριο που θα το, για το τι εστί blockchain και πώς λειτουργεί. Σας παραπέμπουμε και στην ιστοσελίδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Πάντως, είναι σχετικά δύσκολη για παραβίαση η blockchain. Υπάρχει διαφάνεια και τα, ε, τα smart contracts, αυτές οι έξυπνες συμβάσει μπορούν ταυτόχρονα να εκτελούν συμφωνίες πολλών συμβαλωμένων μέρων. Αυτά είναι τα θετικά. Τώρα λιγότερο θετικά, δυσκολίες στην επεκτασιμότητα, μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, θέματα προστασία δεδομένων και άλλες ε, προκλήσεις. Καταρχήν, έχουμε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τις τάσεις που παρουσιάζει και η έκθεσή μας. Βλέπουμε ε, αυξανόμενα μερίδια και πόσα αποφιερώνονται στις τεχνολογίες blockchain. Μάλιστα, όταν συγκεντρώσουμε και άλλα στοιχεία, θα κάνουμε ενημέρωση της έκθεσης. Τρεις τομείς ε, εξετάσαμε για γενικές ε, ε, ευκαιρίες και προκλήσεις. Μία σύντομη επισκόπηση για τις ευκαιρίες στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Χάρη στο blockchain έχουμε εναλλακτικές μορφές νομίσματος, χωρίς την ανάγκη κεντρικής αρχής και σε υποομάδες έχουμε και τις διασυνοριακές ε, πληρωμές που μπορούν να, να γίνονται και μάλιστα σε real time, ε, με real time ενημέρωση και, και επικαιροποίηση. Βέβαια, Έχουμε ακόμη μεγάλη αστάθεια των τιμών και κερδοσκοπία στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Έχουμε κάπως, κάποιους στεναπούς και κανονιστικούς και πρόβλημα στην ε, κανονιστική ρύθμιση για τα ψηφιακά νομίσματα, τα κρυπτονομίσματα. Σε ό,τι αφορά τις ε, αγορές, έχουμε καταρχήν ε, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την έξυπνη κατασκευή και την έχουμε κάποιες ε, πλασματικές, κάποια πλασματικά σενάρια με 250 πλεκόμενους φορείς και η blockchain είναι ένα μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλο παράδειγμα που αφορά τις δημιουργικές βιομηχανίες και το ψηφιακό περιεχόμενο. Το θέμα είναι, ε, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε κουτσομπολιά για παράδειγμα και να τα επαληθεύσουμε για μια συγκεκριμένη ε, γειτονιά. Αυτό είναι το gossip ε, chain, το σενάριο του blockchain που αναπτύξαμε. Επίσης, είδαμε και τα γενικά ωφέλη του blockchain. Καταρχήν, διευκολύνει την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα των συναλλαγών και επίσης ε, εξε, εξασφαλίζει χνηλασιμότητα και εξασφάλιση της προέλευσης. Επίσης, Έχουμε προβλήματα δικαιοδοσιών για αποκεντρωμένα δίκτυα, έλλειψη σαφών κανόνων και ορισμών για τα ε, smart contracts. Επίσης, ε, τι γίνεται με το δημόσιο τομέα και επίσης ευκαιρίες. Έχουμε ε, ακυρότητα των δεδομένων, μη παραβίαση όπως όμως και σε άλλους τομείς βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Πώς μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα συγκεκριμένα πρότυπα ταυτοποίησης μέσα σε συγκεκριμένα συστήματα. Πρέπει να δούμε πώς ο δημόσιος τομέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό προκειμένου να καταφέρει να αυξήσει την συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δηλαδή. Στο τέλος της παρουσίασης αυτής ήθελα να σας δώσω 11 βασικά μηνύματα, δεν τα έχω βάλει με κάποια σειρά προτεραιότητος. Και σας δίνω επίση και κάποιες καταλεκτικές ημερομηνίε τόσο στην έκθεση όσο όμως και στην, στην ιστοσελίδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίε αυτές. Βλέπετε επίσης ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε καταρχάς εφαρμογές όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό οικοσύστημα, τη χρησιμοποίηση ενός μοντέλου blockchain το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία λύση, μόνο ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή, αντιμετώπιση εμποδίων στην όλη διαδικασία της τεχνολογίας αυτής, η έννοια της εμπιστοσύνης και της ε, αποδιαμεσολάβησης. Θα λέγω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη παράνοια. Η τεχνολογία blockchain δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθόλου ενδιάμεση, ότι τους έχουμε εξαλείψει εντελώς δηλαδή. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι, κάποιοι νέοι ενδιάμεσοι να εμφανιστούν στα πλαίσια της τεχνολογίας blockchain. Για παράδειγμα θα μπορούσαν αυτοί να εγγυηθούν την ισότιμη συμβολή στο σύστημα αυτό, την ισότιμη συμμετοχή στο σύστημα και οι νέοι αυτοί ενδιάμεσοι θα μπορούσαν επίσης να εγγυηθούν όσον αφορά την αξιοπιστία. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Όλοι λένε ότι η τεχνολογία blockchain θα δημιουργήσει σε πλήρη αποδιαμεσολάβηση. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ενδεχομένω, όπω σα είπα, να προκύψουν νέοι ενδιάμεσοι. Επίση, θα πρέπει να προκύψει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και κατευντήρες γραμμέ. Θα πρέπει να καταφέρουμε επίση να έχουμε νέε ε, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και τέλος βλέπετε εδώ πέρα ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα παρακολούθησης όπου θα πρέπει εδώ πέρα να έχουμε και μια προορατική στάση. Το σημαντικό είναι να μην παρακολουθούμε μόνο αυτά που συμβαίνουν τώρα αλλά να μπορέσουμε κάπως να προβλέψουμε και να παρακολουθήσουμε αυτά που μας περιμένουν στο μέλλον. Να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες ικανότητες γι' αυτό δηλαδή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ακούσουμε τώρα την επόμενη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα το απόγευμα εδώ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια θέματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά, αν θέλετε, μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όλοι μιλάνε για την τεχνητή ε, νοημοσύνη, αλλά αυτό που έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία οικογένεια μεθόδων, ε, και τεχνολογιών, αλλά υπάρχει ε, μια ολόκληρη ομάδα τεχνολογιών. Μία εξ αυτών είναι το blockchain, μία άλλη ομάδα είναι το ίντερνετ των πραγμάτων το 3D printing, ε, διαφορετικές ε, μορφές ε, υπολογισμού. Όλα αυτά δείχνουν ότι αλλάζει η ζωή μας και γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για ψηφιακή αλλαγή γιατί επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε κοινωνικά σε επαφή, δουλεύουμε, μελετάμε, ταξιδεύουμε. Όλες δηλαδή τις, όλες οι πτυχές της ζωής μας επηρεάζονται από την ψηφιακή αλλαγή. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη, αν θέλει κανείς να πει κάποια βασικά στοιχεία, πρόκειται για το εξή. Γνωρίζετε όλοι σα ότι υπάρχει μια σημαντική γεωπολιτική διαμάχη ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Κίνα για την επικυριαρχία τη τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα έχει επενδύσει ουσιαστικά στην τεχνητή νοημοσύνη και αλλάζει το παραγωγικό τη μοντέλο. Πορά από τα προϊόντα που παράγονταν πολύ φτηνά τώρα πρόκειται να είναι προϊόντα με πολύ μεγάλη αξία. Και γι' αυτό η Κίνα επενδύει στο 5G, σε πολλές τεχνολογίες και κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη. Και βεβαίως οι Ηνωμένε Πολιτείε επικυριαρχούν κυρίως στις εμπορικές εταιρείε. Νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε τη διαμάχη για την Huawei έτσι σαν παράδειγμα για τον ανταγωνισμό, ο οποίος διαδραμαστεί κυρίως σχετικά με την ιδιοκτησία των δεδομένων. Γιατί, διότι σε μεγάλο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ακριβώς γιατί έχουμε μεγάλο όγκο δεδομένων και αναπτύσσεται βέβαια μόνο αν έχουμε αυτό τον όγκο των δεδομένων που επιτρέπει την ανάπτυξη αλγορίθμων. Ω εκ τούτου, η ιδιοκτησία εισαγωγικά, ο έλεγχο, η πρόσβαση στα δεδομένα είναι καθοριστική σημασία. Στην Κίνα, το κράτο ελέγχει όλα τα δεδομένα. Ελέγχει και τα προσωπικά δεδομένα και τα πρόσωπα των οκτώ εκατομμυρίων, 800 εκατομμυρίων χρηστών. Γι' αυτό λοιπόν η Κίνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει αυτή την ε, τεχνολογία αναγνώριση προσώπου ε, και έτσι μπορεί να προχωρήσει και περαιτέρω στους αλγόριθμους. Οι εμπορικές εταιρείες των ΗΠΑ έχουν στην κατοχή τους ε, όλα τα υπόλοιπα δεδομένα γιατί εμείς τους τα δίδουμε. Το 80% 7% όλων των αναζητήσεων περνά από την Google. Όλες οι κοινωνικέ πλατφόρμες είναι αμερικανικέ. και ως εκ τούτου όχι μόνο τους δίνουμε δεδομένα αλλά και τους λέμε γιατί τα δεδομένα είναι σημαντικά. Δίνουμε ένα πλαίσιο για τα δεδομένα και εκεί μέσα να μπορούν να απτύξουν αλγορίθμους. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι μέσα σε όλα αυτά η Ευρώπη προσπαθεί να βρει το δικό τη ε, βηματισμό ε, όχι το κινέζικο μοντέλο, ούτε και το αμερικανικό καθαρά εμπορικό. Η Ευρώπη προσπαθεί ε, να βρει κάποιο ηθικό, ε, ανθρωποκεντρικό μοντέλο, το οποίο προβάλλει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κοινό κέντρο ερευνών, έχει το νέο κέντρο ερευνών, έχει κάνει έρευνες και βλέπετε έχουμε συστήσει μια έκθεση για την τεχνητή νομοσύνη η οποία προσπαθεί να προσφέρει ε, μια πιο σφαιρική εικόνα ε, για τα δεδομένα, το ηθικό στοιχείο, το κοινωνικό, την αντίσταση της κοινωνίας και προσπαθούμε να τα προσφέρουμε όλα αυτά ως μια τροφή εισαγωγικά στους συναδέλφους που δουλεύουν για να καταρτήσουν μια πολιτική και αυτοί δίνουν τροφή περαιτέρω ε, στο συντονισμένο σχέδιο τεχνητής νομοσύνης εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2018. Αυτό το συντονισμένο ε, πρόγραμμα προβλέπει το συντονισμένη δράση όλων των κρατών, γιατί κανεί δεν μπορεί να τα απεξέλθει μόνος του στι ε, προκλήσει και προβλέπει επενδύσει μέχρι και σε 20 δι ευρώ. Προβλέπει επίσης και μια λειτουργία που θα ελέγχει τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν τα κράτη-μέλη. Ε, προβλέπεται επίσης η απορρόφηση και οι επιπτώσεις από αυτές τις επενδύσεις. Εμείς στο κέντρο μας έχουμε ένα iWatch, είναι μια υπηρεσία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνδυασμό με τη Γενική Διεύθυνση ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Εγώ θα σας δώσω έτσι μια ιδέα του τι κάνουμε. Εξετάζουμε το παγκόσμιο σκηνικό. Εδώ βλέπετε την ε, επικυριαρχία των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα παικτών. Έχουμε περίπου 35.000 σημαντικούς ε, παίκτες στην έρευνα ε, και στον εμπορικό τομέα, εταιρείε δηλαδή οι οποίες ασχολούνται με την πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και βλέπετε την κλίμακα των τριών μπλοκ. Οι κόκκινες κουκίδες δείχνουν τον αριθμό των παικτών ε, διερουμένου του συνολικού του αριθμού ε, δια του ΑΕΠ. Ε, και βλέπουμε τις χώρες οι οποίες προχωράνε πολύ περισσότερο. Στην Ευρώπη και πάλι βλέπουμε την ε, κατανομή των χωρών. Έχουμε χώρες οι οποίες ε, ε, έχουν υιοθετήσει το, την τεχνητή νομοσύνη. Σημαντική χώρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και το ότι έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Στο επόμενο θεματική εξειδίκευση στην Ευρώπη είμαστε πολύ εξειδικευμένοι σε γενικές υπηρεσίες και στη ρομποτική και επίσης ε, και ε, στις μπλε περιοχές στα CAVs, ε, Connected to All Vehicles. Στην Κίνα, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πολύ ισχυρή στην αναγνώριση προσώπου. Η ρομποτική είναι πολύ σημαντική στην Ευρώπη. Είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή, αλλά και η σημαντικότερη εξαγωγή. Έχουμε μια ιδιαίτερα ανοιχτή οικονομία και αυτό είναι σημαντικό. Η Κίνα όμω πρόσφατα μα ξεπέρασε ε, είναι ο πιο σημαντικός ε, παραγωγός, ε, αλλά κυρίως εξυπηρετεί την εσωτερική της αγορά. Στην έρευνα και την ανάπτυξη βλέπετε και πάλι την κατανομή αναχώρες, βλέπετε τους βασικούς παίκτες, τον κόσμο. Η Ευρώπη και πάλι βρίσκεται σε καλή θέση, τουλάχιστον για την τεχνολογία εχμής. Εξετάζουμε την τεχνητή νομοσύνη και στις δημόσιες υπηρεσίες. Έχουμε συγκεντρώσει πολλές μελέτες και θέλω να σας πω ότι οι δημόσιες υπηρεσίες όλες κάνουν πειράματα με την τεχνητή νομοσύνη, αλλά δεν έχουν καταφέρει και πάρα πολλά. Συμπέρασμα, ε, η τεχνητή νομοσύνη είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η Ευρώπη έχει πολλές ευκαιρίες στον διεθνή ανταγωνισμό, έχει καλή έρευνα, έχει μια πολύ καλή πολιτισμική ποικιλομορφία. Σε μεγάλο βαθμό πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας. Ως εκ τούτου το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι ότι το μέλλον εξαρτάται από εμά. Ε, Εμεί θα το χαράξουμε και θα το διαμορφώσουμε και αν δεν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος. Περνάμε τώρα στους συντονιστές κύριε Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο παρουσιάσεις. Συνοψίσατε ουσιαστικά τις μείζονε προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο εγγύς μέλλον. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να μείνουμε πίσω σε αυτό τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, σε αυτή την τεχνολογική επανάσταση. Και είπατε εύστοχα ότι έχουμε πολύ προηγμένη έρευνα και έχουμε και ένα πάγιο κανονιστικό πλαίσιο αλλά και οδοντολογικό και γενικώ κάνουμε πολλέ προσπάθειε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ και ειδικότερα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, έχουμε πολύ σημαντικέ ε, εταιρείε που ε, πρωτοστατούν στην παγκόσμια αγορά. Πάντως, η ιστορία και στο παρελθόν μας έχει διδάξει ότι Ακόμη και με όλα αυτά τα θετικά συστατικά που έχουμε, δεν καταφέρουμε στην Ευρώπη να κρατήσουμε την υπεροχή μας και την ηγετικό μας ρόλο. Και αναφερθήκατε σε κάτι που είναι αρκετά ανησυχητικό. Μιλήσατε για τις πλατφόρμες που απαιτούνται και που δεν είναι ευρωπαϊκές. Οπότε, τι συμβουλή έχετε να μας δώσετε για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πώς να μεριμνήσουμε ώστε αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε πίσω και δεν θα χάσουμε την ηγετική μας θέση. Και η τεχνολογία της πέμπτης γενιάς τηλεπικοινωνιών θα σημάνει ένα σημαντικό μετασχηματισμό και για την κοινωνία και για τη βιομηχανία μας και θα καταφέρουμε να κρατήσουμε την τεχνολογική μας ηγετική θέση. Κάτι που δεν καταφέραμε πάντα στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Κυρία Τόγια από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή. Άκουσα το τελευταίο τμήμα της παρουσίασής σας, την πρώτη την άκουσα μέσω του web streaming. Όντω, από το, κέντρο, το κοινό κέντρο ερευνών πάντα έχουμε πολύ σημαντικέ ενδείξει και πολύ σημαντικά δεδομένα για μα που καλούμεθα να χαράξουμε πολιτική και να λάβουμε αποφάσει. Πολύ σημαντικά το όσα μα είπατε, ιδίω ένα πεδίο το οποίο εξελίσσεται συνεχώ. Σήμερα το πρωί ήμουνα στο δικό μου το κράτο μέλο, στην Ιταλία, στη Λομβαρδία συγκεκριμένα και ορισμένοι σήμερα το πρωί μου μιλούσαν ακριβώ για την εργασία που κάνετε εσεί στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο του κέντρου ερευνών. Λοιπόν, έχω να κάνω μία ερώτηση. Πολύ σωστά είπε η συνάδελφο, πώ μπορούμε να διατηρήσουμε την τεχνολογική μα κυριαρχία με το 5G και τα άλλα δίκτυα. Εγώ να κάνω ένα ακόμα ερώτημα παρεμφερέ. Πώ μπορούμε να διατηρήσουμε τη δική μα την κυριαρχία, αν θέλετε, και ικανότητα την επιχειρηματική. Πριν από λίγο είπατε ότι είμαστε στη ρομποτική για παράδειγμα στην πρώτη θέση και ξέρω ότι για παράδειγμα έχουμε και μια πολύ σημαντική μεταποιητική βιομηχανία και μια βιομηχανία παραγωγής μηχανών. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς βάσει της δικής σας της μελέτης, την οποία θα διαβάσω πολύ προσεκτικά, να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη πέρα από την τεχνολογική κυριαρχία θα καταφέρει να κρατήσει και την βιομηχανική και παραγωγική της κυριαρχία. Σας ευχαριστώ. For ε, Europe is anybody Είναι κανείς από την ομάδα Renew Europe? Όχι, οπότε πάμε στους πράσινους. Ο κύριος Νίνιστο. Σας ευχαριστώ. Ε, κάνετε κάποιες φιλο, φιλοσοφικές σκέψεις για το πόσο μπορούμε να έχουμε το προβάδισμα στην Ευρώπη για την τεχνητή νοημοσύνη και την ε, πέμπτη γενιά τηλεπικοινωνιών ε, στο παρελθόν έχουμε, είχαμε καταλήξει σε κάποια θεμελιώδη στοιχεία που είναι σημαντικά, αλλά ακόμη δυστυχώς προηγούνται οι Αμερικανοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν να πάρουμε κάποια μαθήματα ίσως και από αυτούς και για την πέμπτη γενιά των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Σίγουρα έχουμε ευρύτατες γνώσεις, αλλά πώς ε, θα μπορέσουμε το οικοσύστημα, το επιχειρηματικό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το εξάγουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή το εμπορικό σκέλος να αναπτύξουμε. Να μην παραμείνει εσωτερικό θέμα αυτό. Ε, να έχουμε ηγετικό ρόλο και παγκοσμίω σε θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και τις γνώσεις που έχουμε στους τομείς αυτούς, ίσως θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τα θέματα ενεργειακής, ενεργειακών προτύπων και οικονομίας με την Πράσινη Συμφωνία και σίγουρα η ενεργειακός μετασχηματισμός συμπεριλαμβάνει και την ψηφιοποίηση. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για την ενεργειακή απόδοση και ε, είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά τέτοια θέματα, ιδιαίτερα στη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων. Πώς λοιπόν θα προωθήσουμε τα θέματα αυτά τα περιβαλλοντικά, ώστε να ενισχύσουν και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν από την ταυτότητα και δημοκρατία. Περνούμε στο, στην ομάδα ECR. Εγώ συντονιστή, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να υποβάλω κάποιε ερωτήσει, γιατί ο αναπληρωτή συντονιστή απουσιάζει. Μία γενική παρατήρηση πρώτα θα ήθελα να κάνω. Μιλήσατε για τον ευρωπαϊκό τρόπο, τον τρίτο τρόπο δράσης. Εγώ θυμάμαι τότε που μιλούσαμε για την αντιπαλότητα των δύο συστημάτων του Αμερικανικού και του Κινέζικου και είπαμε ότι ίσως χρειάζεται ένας τρίτος δρόμος. Ο τρίτος δρόμος όμως μπορεί να είναι και ουτοπικός, να είναι μια ψευδέστηση. Θα μπορούσατε εσείς να μας προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά που θα έχει ένας τέτοιος τρίτος δρόμος ε, μεταξύ του ιδιωτικού κλάδου που προσανατολίζεται προς την αγορά, που είναι το ένα μοντέλο και το άλλο μοντέλο είναι ε, η δημόσιο, το, ο κρατικός ε, παράγοντας που είναι ο πιο ισχυρός και καθορίζει και καθοδηγεί την όλη διαδικασία. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων, πώς βλέπετε τον τρίτο δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία και το δυναμικό που έχει η Ευρώπη, ειδικά τώρα και μετά το Brexit, ε, παρόλο που αποχώρησε ένας πολύ σημαντικό εταίρος μας στα θέματα αυτά, αυτό που μας ε, προβληματίζει είναι πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό του συνόλου της Ευρώπης. Γιατί το ευρωπαϊκό σχέδιο ανέκαθεν προσπαθούσε να βρει μια ισορροπία στην ανάπτυξη. Αλλά και στην ψηφιακή βιομηχανία και στον ψηφιακό κλάδο θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που δεν θα είναι ε, μόνο σε ένα ίδιο κέντρα, αλλά θα αξιοποιούν το δυναμικό του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το blockchain και την ενέργεια, είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί το, οι τεχνολογίες blockchain είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Θα μπορούσατε όμως να μας εξηγήσετε πιο διεξοδικά πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και αν υπάρχουν και οι σκοτεινές πλευρές ε, της τεχνολογίας blockchain ως προς τα ενεργειακά θέματα. Ε, ε, αν οι συναλλαγές μέσω τεχνολογιών blockchain αφήνουν ένα αποτύπωμα άνθρακα πολύ μεγαλύτερο από ότι ε, η σημερινή τρόπη συναλλαγών. Άλλος κανείς δεν βλέπω να ζητά το λόγο, οπότε από τους συντονιστές, οπότε περνάμε στους υπόλοιπους. Ε, κύριε Σπυράκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Έχω να κάνω κάποιες ουσιαστικές ερωτήσεις, αλλά μερικές φορές νομίζω ότι για τα ζητήματα αυτά χρειαζόμαστε και περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχάς, πόσα χρήματα, πόσες επενδύσεις χρειαζόμαστε προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να έχουμε ένα ανταγωνιστικό κλάδο τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε την ηγετική θέση της Κίνας ή μια αναδυόμενη ηγετική θέση επίσης από τις ΗΠΑ και εμείς είμαστε απλώς μέρος, αν θέλετε, του παιχνιδιού αυτού. Έχουμε την Ericsson και την Nokia, τις δύο μόνο αυτές επιχειρήσεις που εμπλέκονται είναι τελικά οι μόνες ή έχουμε κάτι παραπάνω. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο και πιο δυναμικά. Η δεύτερη ερώτηση. Θεωρείτε πραγματικά ότι όσον αφορά τη ρύθμιση, τους κανονισμούς, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τα κρυπτονομίσματα. Πολύ φοβάμαι ότι ο τομέα των κρυπτονομισμάτων θα εξελίσσεται και θα μετασχηματίζεται πολύ γρηγορότερα από ότι εμεί θα καταφέρνουμε να νομοθετούμε στον τομέα αυτό και στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών. Ο κύριο Πεκάρινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Η τεχνητή νοημοσύνη για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι εξαρτάται πάρα πολύ και από το τι πρόοδο εμείς θα καταφέρουμε να πετύχουμε στο πλαίσιο του τομέα 5G, καθώς επίσης και σε άλλους τομείς υπολογιστικής. Ξέρω ήδη ότι οι ορισμένε χώρες έχουν γίνει πολύ σημαντικά άλματα έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος ακόμα και στην τεχνολογία 6G. Τα δύο αυτά ζήματα λοιπόν, το 5G και η κβαντική υπολογιστική, πόσο θα επηρεάσουν τελικά τη θέση μας σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί την κβαντική υπολογιστική που την έχουν στις ΗΠΑ στην Κίνα, εμείς δεν τη διαθέτουμε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο σημαντικοί λοιπόν οι παράγοντες αυτοί. κύριο Σκοτουόρθι. Όχι, δεν θέλετε το λόγο που τη βλέπω. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Gracias. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους εμπειρογνώμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών για την εξασφάλιση της ασφάλισης των δικτύων 5G και τη δυνατότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν επιθέσεις που μπορούν να απειλήσουν διάφορους τομείς της ζωής μας, γιατί οι μελλοντικέ τηλεπικοινωνίες θα είναι πανταχού παρούσες. Οπότε χαίρομαι που τονίζετε την ανάγκη συντονισμού. Πάντως, στα θέματα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν να υιοθετήσουν μέτρα και να εξασφαλίσουν αρμοδιότητε στι ρυθμιστικές αρχέ για να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα του κινδύνου. Ήδη στην έκθεση του Οκτωβρίου είχαμε εντοπίσει κάποιου κινδύνου και τώρα τα συμπεράσματα λένε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν κάποια μέτρα. Ποια είναι η κατάσταση ασφάλεια που έχουμε σήμερα, σε τι κατάσταση τιμότητα βρισκόμαστε, έχουν θεσπιστεί κάποια μέτρα και πώ θα εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα τη εσωτερική αγορά αν ένα κράτο αποφασίσει να αποκλείσει μια επιχείρηση, ένα άλλο κράτος δεν θα την αποκλείσει. Τέλος, ε, θα προωθηθούν κάποια συστήματα, ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης. Ευχαριστώ. Um, δεν βλέπω άλλου συναδέλφου να ζητούν το λόγο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στου καλεσμένου εμπειρογνώμονέ μα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για να απαντήσουν σε απορίε των συναδέλφων και να καταλήξουν ενδεχομένω και σε κάποια συμπεράσματα. Όντως, πολλές ερωτήσεις ε, αφορούσαν το ίδιο θέμα, γι' αυτό θα τις ομοδοποιήσω. Και αν ε, ε, μερικοί δεν μείνουν ικανοποιημένοι από την απάντηση, που σίγουρα θα ισχύει αυτό, μπορούν να επανέλθουν. Υπάρχει σαφώς το θέμα του να εξασφαλίσουμε και να διατηρήσουμε το προβάδισμα σε θέματα ρομποτικής, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και να διασφαλίσουμε τον ηγετικό μας ρόλο βρίσκοντας το δικό μας τρόπο δράσης. Και όταν μιλούμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλούμε για μεθόδους που είναι 40, 50, 60 χρόνων. Αλλά αυτό που άλλαξε την τελευταία επταετία κυρίω είναι ο όγκος των δεδομένων και ο όγκος της επεξεργασίας τους. Ε, εκεί έγκυται το ποιοτικό άλμα των τελευταίων χρόνων. Και σίγουρα η στρατηγική μας θα πρέπει ε, να είναι πολυεπίπεδη και πολυσχηδής. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο σε μία μόνο λύση. Θέλουμε καταρχήν καλύτερο έλεγχο των ευρωπαϊκών δεδομένων και καλύτερη χρήση των δεδομένων που έχουμε στην Ευρώπη και αύξηση της ικανότητα επεξεργασίας των δεδομένων μας στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Άλλο θέμα που συνδέεται και με το ζήτημα των τηλεπικοινωνιών πέμπτη Γενιά είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψη η αλλαγή του μοντέλου. Μέχρι στιγμής είχαμε κυρίως ε, όλο και περισσότερα δεδομένα, αύξηση του αριθμού των δεδομένων που ε, συγκεντρώνονταν σε εκτεταμένες υποδομές. Τώρα όμως όσο έχουμε όλο και περισσότερες αισθητήρες, δίκτυα αισθητήρων και το διαδίκτυο των πραγμάτων, το πρότυπο θα αλλάξει. Και αντί να έχουμε κέντρα επεξεργασίας δεδομένων ε, που θα συγκεντρώνουν τα δεδομένα, θα έχουμε όλο και περισσότερο επεξεργασία των δεδομένων που θα γίνει στις παρυφές του δικτύου, στους αισθητήρε, όπως ε, τα κινητά, για παράδειγμα, που ήδη έχουν, κάνουν μεγάλο τμήμα της επεξεργασίας. Οπότε θα έχουμε στους δορυφόρους, στους αισθητήρε παρυφές του δικτύου την επεξεργασία και θα μεταφέρουμε πολύ λιγότερα δεδομένα μέσα στο δίκτυο. Και αυτή η αλλαγή του, του προτύπου, του τρόπου σκέψης θα τροποποίησει τη σημερινή κατάσταση και σε σχέση με τι πλατφόρμε. Οι πλατφόρμε σήμερα έχουν ισχύ γιατί συγκεντρώνουν ε, όλα αυτά τα δεδομένα και όσο περισσότερα δεδομένα έχουν τόσο μεγαλύτερη ισχύ του είναι. Τώρα, αν αλλάξουμε αυτό τον τρόπο σκέψη, θα δημιουργηθεί χώρο και ε, θέση που μπορούμε εμεί να τη διεκδικήσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει αυτή την ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε. Σίγουρα ο συνάδελφο θα αναπτύξει περισσότερο το θέμα τη πέμπτη γενιά τηλεπικοινωνιών και τη ε, κυβερνοασφάλεια. αλλά Σίγουρα μόνο με συνεργασία θα έχουμε ευκαιρία εν τη ενός Όσο περισσότερο κατακαιρματισμένοι είμαστε, τόσο πιο αποδυναμωμένοι θα γίνουμε. Και τόσο πιο μικρό θα είναι το μερίδιό μας. Και πολύ σωστά ε, επισημάνατε την ανάγκη συνεργασίας. Και για την τεχνολογία blockchain το αφήνω στο συνάδελφο. Και το θέμα της πέμπτης γενιάς τηλεπικοινωνιών συνδέεται με τη μετάβαση προς το ίντερνετ των πραγμάτων και την αύξηση της επεξεργασίας των δεδομένων στις παρυφές του δικτύου και όχι τόσο σε κέντρα δεδομένων. Οπότε θα αλλάξει το μοντέλο πια. Αυτά και θα δώσω, θα αφήσω τα υπόλοιπα στον Αλεξάνδρ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όχι μόνο για το θέμα της ε, τεχ, ε, σε θέματα ενέργειας, αλλά και γενικότερα το πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε την κυριαρχία μας σε πολλούς τομείς. Στο blockchain, κοιτάξτε, αυτή η μελέτη περιλαμβάνει άλλη μία που αφορά θέματα βιομηχανίας. Για το blockchain, μία από τις μεγάλες προκλήσεις, που δεν είναι βέβαια καινούργια, γιατί η τεχνολογία του blockchain υπάρχει εδώ και 50-60 χρόνια. Απλά τώρα βλέπουμε σε συμπυκνωμένη μορφή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα unicorn, και ε, ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι παίκτες που θα εργαστούν με διαφορετική ταχύτητα. Η Ευρώπη δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε όπου αν αποτύχει μια μεγάλη αγορά ε, τότε θα εμφανιστεί σε μια άλλη αγορά. Στην Ευρώπη δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα δηλαδή αυτό που είδαμε πρόσφατα στο blockchain είναι ότι έχουμε μικρές ε, εταιρείε οι οποίες θα είναι κρίσιμη μάζα για το μέλλον. Και αυτό ισχύει και για την πέμπτη γενιά τηλεπικοινωνιών. Ω εκ τούτου, ένα από τα βασικά θέματα που τώρα η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει είναι το πώς μπορεί να συμπεριλάμβει το blockchain, την κβαντική υπολογιστική, ε, την τεχνητή νομοσύνη, όλα αυτά, όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες Αυτά, όπως σας είπα, υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό ε, στην παραγωγή. Υπάρχουν τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα, δηλαδή, αυτά που υπάρχουν απλά είναι να τα βάλουμε στην κορυφή. Το blockchain και την τεχνητή νομοσία. Να δώσουμε την πρώτη προτεραιότητα. Αυτή η ιδέα του τρίτου τρόπου και αυτό είναι δύσκολο, γιατί ακούμε ε, εδώ και αρκετέ δεκαετίες για ένα εναλλακτικό τρίτο τρόπο. Ακούμε για εναλλακτικό τρίτο τρόπο για την τεχνολογία. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει από τις έρευνές μας είναι ότι είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε αυτό στην Ευρώπη. Εμείς όμως έχουμε αξίες και κανονισμούς που αυτή τη στιγμή λειτουργούν και κανονισμούς που μπορούν να λειτουργήσουν προορατικά για το μέλλον. Ως εκ τούτου προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο με βάση ηθικές αξίες. Τώρα, το τι σημαίνει ηθικές αξίες, αυτό μπορεί να συζητηθεί, αλλά είναι κάτι που το ευρωπαϊκό σύστημα των τεχνολογιών, ακόμα και το παλιό σύστημα, προσπαθεί να το προβάλλει. Τώρα, τα κρυπτονομίσματα και οι κανονισμοί. Είναι δύσκολο να παρακολουθεί κανείς όλα τα κρυπτονομίσματα και τους κανονισμούς. Από τις έρευνες μας διαπιστώσαμε ότι η Ευρώπη μπορεί να προβλέψει όσο το δυνατόν περισσότερα, να εντοπίσει ε, το τι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Ε, token, κρυπτοκεφάλαια, αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ε, κανονισμούς στο μέλλον. Δύσκολο, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να συντάσσουμε κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικούς κανονισμούς και αυτέ οι ε, καθευθυντές μας μπορούν να περνάνε την κατηγοροποίηση των κεφαλαίων. Ε, το τι είναι εκτός και τι εντός των ε, κανονισμών και το τελευταίο blockchain στην ενέργεια. Το blockchain έχει αυτό το δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή από τη μια όλοι μιλάνε για το blockchain ε, που καταναλώνει χώρο και είναι αλήθεια. Όμως τα νέα πρωτόκολλα του blockchain δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μείωση τουλάχιστον τα πρωτόκολλα που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη το blockchain μας δίνει και νέες σκέψεις για smart grids, εφή, δίκτυα ε, χρησιμοποιώντας ε, με ευφυή τρόπο, δύσκολο και αυτό να το ορίσουμε, αλλά το blockchain κατά κάποιον τρόπο με ευφυή συμβάσεις αυτοματοποιεί τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα ευφυή δίκτυα στις ε, διαπραγματεύσεις για την ενέργεια και στο ενιαίο ερευνητικό κέντρο ασχολούμεθα και με τις ε, ε, αγορές ενέργειας, Καινούργιο αυτό είναι το blockchain, όπου τις συμβάσεις δεν θα τις διαπραγματεύονται άτομα, αλλά τεχνητές μονάδες Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι το blockchain είναι κακό για το περιβάλλον, αλλά υπάρχει και άλλοι που λένε ότι μπορούμε με το blockchain να κερδίσουμε σε ενέργεια. Ακούστηκε επίσης και μία ερώτηση για το πώς θα τα καταφέρουμε. Και δεν τα καταφέραμε πολύ καλά στο παρελθόν. Πάλι εδώ πέρα έχουμε ένα συνδυασμό, αν θέλετε, ανάμεσα στο ότι πάρα πολλές από αυτές τις τεχνολογίες έχουν να κάνουν με την έννοια της εμπιστοσύνης και η εμπιστοσύνη είναι σημαντικότατη παγκοσμίω. Είναι σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται η εμπιστοσύνη. Αυτό πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστικό. Για παράδειγμα, με το GDPR. Από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί αντιγράφουν το δικό μας το μοντέλο. Η Καλιφόρνια, για παράδειγμα, έχει εγκρίνει μια νομοθεσία που συνάδει πάρα πολύ με το GDPR και ο κύριο Ζούκεμπερκ μιλώντα στο Κογκρέσο, το Αμερικανικό, είπε ότι ενδεχομένω εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα πήγε καλά. Ενώ ξέρετε ότι αρχικά είχαμε δεχθεί πάρα πολλέ επικρίσει για το GDPR, τον Γενικό Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων. Θεωρώ ότι εναπόκειται σε εμά και έχουμε πραγματικά πολλέ σημαντικέ ευκαιρίε. Η κυρία Τόη αναφέρθηκε στις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε στο πλαίσιο της μεταποίησης της βιομηχανίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα ωφελήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πολύ ενδιαφέρουσε και οι δύο παρουσιάσεις. Καταδείξτε πραγματικά ότι είναι αμφίσιμε πολύ συνήθω οι τεχνολογίες και ότι τίθεται πάντα και το ζήτημα των κανονισμών, καθώς επίσης και οι κοινωνικές και οικονομικές πτυχές τη ρύθμιση αυτή. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ και σίγουρα τα ζητήματα αυτά θα μας απασχολήσουν πολλέ φορέ και στο μέλλον. Σα ευχαριστούμε. Περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, όπου έχουμε εδώ ανακοίνωση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όσον αφορά την ασφαλή εγκατάσταση του 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω ολόθερμα τον κύριο Μιγγέλ Γκονζάλε Σάντσο Μποτέρο, επικεφαλή τη Μονάδα Τεχνολογία Κυβερνοασφάλεια και Οικοδόμηση Ικανοτήτων από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων και Περιεχομένου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία ώρα μπορούμε να διαθέσουμε σε αυτό το σημείο. Και για μία ακόμη φορά θα ήθελα να μας πείτε αν θέλετε να λάβετε το λόγο συζήτηση αυτή, σηκώντα το καρτελάκι σας και να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα για την παρουσίασή σα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την εργαλειοθήκη για την κυβερνοασφάλεια στη στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 5 γενιάς. Έχω και διαφάνειες μαζί μου. Εγώ θα κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση της σημασίας που έχει η πέμπτη γενιά των τεχνολογιών ε, κινητών τηλεπικοινωνιών και πώς ε, συνδυάζεται με το θέμα της ασφάλειας. Και θα σας εξηγήσω την πρόσφατη μας δημοσίευση της 29ης Ιανουαρίου, τη λεγόμενη εργαλειοθήκη ε, για τα μέτρα μετρίασης της ασφάλειας για τη 5G και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ίδιο θέμα. Καταρχήν, μια ανακεφαλαίωση. Είναι πραγματικά μια ρηξικέλευτη τεχνολογία η πέμπτη γενιά. Δεν είναι μια αναβάθμιση της προηγούμενης ε, τέταρτης γενιάς ε, των κινητών δικτύων τηλεπικοινωνιών. Η πέμπτη γενιά και η σχετική τεχνολογία θα μεταρρυθμίσει άρτην την οικονομία και την κοινωνία μας. Εξού και οι θερμές συζητήσεις για την ανάπτυξη και την ασφάλεια της πέμπτης γενιάς των δικτύων. Ακριβώς γιατί η σημασία των τεχνολογιών αυτών και η εξάρτηση που θα έχει η οικονομία και η κοινωνία μας από αυτές, αλλά και το γεγονός ότι οι αγορές στην Ευρώπη είναι αλληλοσυνδεόμενες, εξηγούν όλο τον προβληματισμό και τις ανησυχίες για την ασφάλεια αυτής της τεχνολογίας. Γιατί οι επιπτώσεις ασφάλειας ή συμβάντων ασφάλειας τεχνολογίας θα είναι τεράστιες. Και αυτό σχετίζεται και με την ανάπτυξη της, και εξέλιξη της τεχνολογίας που στηρίζεται σε λογισμικό, όπου ναι, η τεχνητή ε, νοημοσύνη θα βρίσκεται στην καρδιά, αλλά και στην περιφέρεια, που δημιουργεί τεράστιε προκλήσεις για την ασφάλεια αυτής της τεχνολογίας και οι μέχρι στιγμής προσεγγίσεις ίσως δεν αρκέσουν στο μέλλον για να εξασφαλιστεί η θωράκιση αυτών των τεχνολογιών. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα της ασφάλειας, ύψιστη προτεραιότητα. Και εδώ έχουμε την ανάπτυξη παρουσίαση των δικτύων πέμπτης γενιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί με αρκετή ταχύτητα στο παγκόσμιο προσκήνιο, με δοκιμές της τεχνολογίας αυτής ε, να εφαρμόζονται παντού στην Ευρώπη. Αλλά βέβαια δεν θα γίνει εν μία νυχτή η πλήρης ανάπτυξη της πέμπτης γενιάς είναι χρονοβόρα διαδικασία, θα χρειαστούν κάποια χρόνια ακόμη. Εξού και η ανάγκη της επίλυσης των ζητημάτων ασφάλειας, γιατί μιλούμε και για πολύ σημαντικές επενδύσεις που προϋποθέτουν μια ασφάλεια για τους φορείς και τους παράγοντες της αγοράς. Πέρυσι είχαμε στη δημόσια συζήτηση το θέμα αυτό της μελλοντική ασφάλειας των δικτύων πέμπτης γενιάς. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγύψει στο ζήτημα αυτό, ήδη το Μάρτιο, κάτι που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπέβαλε μία σύσταση για την οργάνωση των ε, εργασιών για το θέμα της ασφάλειας των δικτύων της πέτης γενιάς και γίνεται κυρίως μέσω της οδηγίας ΝΙΣ, για τις ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Και υπάρχει μάλιστα ε, μία ομάδα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οργανισμού ε, ΕΝΙΣΑ, που είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων. Οπότε γύψαμε στο θέμα της ασφάλειας και καταλήξαμε σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για να διασκεδαστούν οι ανησυχίε μας για την ασφάλεια. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε πέρυσι το Μάρτιο και συνεχίζεται με το έγγραφο για την εργαλειοθήκη. Καταρχήν, τα κράτη-μέλη ε, διενέργησαν τους εθνικούς κινδύνους αξιολόγηση κινδύνου πέρυσι το καλοκαίρι και τον Οκτώβριο είχαμε έναν, μια ευρωπαϊκή συντονισμένη αξιολόγηση κινδύνου με συνενετική βάση για τους κινδύνους των δικτύων της πέμπτης γενιάς και τέλος τον Ιανουάριο, όπως σας είπα, φέτος τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την εργαλειοθήκη των μέτρων μετριασμού των κινδύνων που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση κινδύνου που κάναμε τον Οκτώβριο του 2019. Οπότε αυτή η αξιολόγηση κινδύνου εντόπισε νέα κατηγορίες. Καταρχήν ήταν σημαντικό να συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη ε, επί της μεθοδολογίας για την προσέγγιση και την ανάλυση των προβλημάτων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός ΕΝΙΣΑ ενεπλάκησαν ενεργά στη διαδικασία και εντοπίσαμε πέντε απειλές ε, στα κίνδυνα. Και προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα πιο ευάλωτα και τα τροτά σημεία του συστήματος. Ε, ποια είναι τα πιο ευάλωτα λοιπόν και τώρα τα σημεία και καταλήξαμε σε σενάρια κινδύνου. Δηλαδή, ήδη κινδύνου τεχνικού κινδύνου, όπως τα σφάλματα ρυθμής παραμέτρου δικτύου, η έλλειψη ελέγχων πρόσβασης ή κάποιους ε, παράγοντες απειλής που θα μπορούσαν είναι και κρατικοί παράγοντες, οργανωμένα έγκλημα, εγκληματικές οργανώσεις ε, και ούτω καθεξής. Και τα βασικά πορίσματα ήταν ότι η ασφάλεια της πέμπτης γενιάς ε, αυξάνει το την επιφάνεια του κινδύνου λόγω των εξελίξεων της τεχνολογίας. Έχουμε μια τεχνολογία που εδράζεται περισσότερο στη, ε, στο λογισμικό, στην, ε, στις πληροφορίες, στα, στις παρυφές του δικτύου και κάτι τέτοιο αυξάνει το επίπεδο ανησυχίας ως προς το κίνδυνο. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία ως προς την ανάλυση του κινδύνου. Ε, η ανάλυση λοιπόν του κινδύνου έγινε βάση του κινδύνου και βάσει συνένεση των κρατών μελών. Έτσι εντοπίσαμε τους παράγοντες κινδύνου. Μετά την ε, αξιολόγηση, τη συντονισμένη ευρωπαϊκή αξιολόγηση κινδύνου που στηριζόταν στις εθνικές αξιολογίες κινδύνου, καταλήξαμε στην εργαλειοθήκη που υιοθετήσαμε στις 29 Ιανουαρίου του 2020. Και αυτό δεν ήταν ε, προϊόν της Επιτροπής μόνο. Ήταν ένας καρπός συνεργασίας με τον ΕΝΙΣΑ και με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομάδα συνεργασίας στην οποία συμμετείχαν και τα κράτη-μέλη. Οπότε ήταν μια πολιτικά καθοδηγούμενη διαδικασία βάσει συμφωνία και όχι με την παραδοσιακή μέθοδο τη υποβολή πρώτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ακόλουθε διαπραγματεύσει. Προηγήθηκε μια πολιτική συμφωνία. Οπότε αυτό η εργαλειοθήκη για, το μετριασμό των κινδύνων ουσιαστικά εντοπίζει μη διάφορα μέτρα, στρατηγικά, τεχνικά και υποστηρικτικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Θα σας τα αναφέρω εντάχει. Στη συνέχεια καθορίζουμε σχέδια μετριασμού των κινδύνων Δηλαδή, βασικές κατηγορίες ε, των σενάριων κινδύνου, που είναι εννέα, όπως σας είπα, που εντόπισαν τα κράτη-μέλη. Και για τις εννέα αυτές κατηγορίες ε, εντοπίζουμε κάποια κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Για παράδειγμα, ένα σενάριο κινδύνου είναι η εξάρτηση από ένα και μόνο προμηθευτή για την τεχνολογία. Οπότε τι μέτρα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σενάριο τη εξάρτηση από ένα και μόνο προμηθευτή. Και τέλο και κάποια συμπεράσματα και συστάσει προ τα κράτη-μέλη και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα μέτρα είναι 8 στρατηγικά μέτρα, 11 τεχνικά μέτρα και 10 υποστηρικτικά μέτρα που ενισχύουν ουσιαστικά τις κανονιστικές ε, αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών που επιβλέπουν κυρίως ε, φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων. Έχουμε μέτρα για τους προμηθευτές, το προφίλ κινδύνου των προμηθευτών, τη διαφοροποίηση των προμηθευτών τεχνολογίας, ενίσχυση ικανοτήτων. Αυτά είναι τα στρατηγικά μέτρα και έχουμε και πιο τεχνικά μέτρα που είναι κάποιες βασικές προϋποθέσεις και ειδικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών του εξοπλισμού και ούτω καθεξής. Αυτή η διαφάνεια ουσιαστικά ανακεφαλαιώνει αυτά τα μέτρα, στρατηγικά και τεχνικά και υποστηρικτικά. Και τέλος, για να ολοκληρώσουμε τη μεθοδολογία μας, συνδέουμε αυτά τα μέτρα με τα σενάρια κινδύνου τα εννέα σενάρια κινδύνου που εντοπίσαμε τον Οκτώβριο. Οπότε πρόκειται για περίπλοκους κινδύνους και άρα χρειάζεται ένα συνδυασμός μέτρων για να αντιμετωπιστούν. Βέβαια, οι καταστάσεις μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις εξελίξεις αγοράς και κάποιους άλλους παραμέτρους. Οπότε, εκεί θα γίνει κάποια προσαρμογή στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίσει βάσει της κοινή προσέγγισης, αλλά προσαρμόζοντας τις δικές του συνθήκες. Εδώ είναι ένα παράδειγμα σχεδίου μετριασμού, με το δεύτερο σενάριο κινδύνου, που αφορά τη... το ποιος έχει πρόσβαση στο δίκαιο και κίνδυνος για την πρόσβαση. Και στα αριστερά, στη ΜΟΒ στήλη, έχουμε ενίσχυση κανονιστικών ελέγχων, ενίσχυση του ρόλου των εθνικών αρχών, η διενέργεια ελέγχων και επίση βλέπουμε πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα μέτρα και τι παράμετρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή του. Κάτι που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι τα κράτη-μέλη τα, κρατη ίδια κατέληξαν σε αυτέ τι αξιολογήσει. και αυτά κατά τη γνώμη του είναι τα πιο κατάλληλα μέτρα για συγκεκριμένου κινδύνους και κατέληξαν και σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του. Τώρα, όσον αφορά στα συμπεράσματα από αυτή την εργαλειοθήκη, ε, για τα, τα κράτη-μέλη καλούνται να ενισχύσουν ε, τις προδιαγραφές ασφαλείας σε σχέση με το 5G, να εξετάσουν ε, το προφίλ κινδύνου των προμηθευτών και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να στηρίξει μια διαδικασία μέσα από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Όπως σας είπα λοιπόν και προηγουμένως, αυτό είναι το έγγραφο για τα κράτη-μέλη από την ομάδα συνεργασίας. Ε, το έγγραφο συνοδεύτηκε και από μια ανακοίνωση επιτροπής της ίδιας ημέρας που σε μεγάλο βαθμό ε, επιτυγχάνει τρία πράγματα. Πρώτον, εγκρίνει την εργαλειοθήκη. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πλήρω αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, συστήνει στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ε, κατ' ουσίαν μέχρι τις 30 ε, Απριλίου, να έχουν ληφθεί μέτρα για να εφαρμοστεί η εργαλειοθήκη, για να διατηρηθεί ο δυναμισμό. Και το τρίτο πράγμα που κάνει η ανακοίνωση είναι να υπενθυμίσει ότι υπάρχουν εργαλεία ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν μέτρα εξασφάλισης ε, που μπορούν να στηρίξουν και την καινοτομία. Βεβαίω, ε, κανόνε για τι τηλεπικοινωνίε, για την κυβερνοασφάλεια, αυτά υπάρχουν σήμερα και ε, έτσι μπορεί να μπορούν να προβλεφτούν κάποιες δεσμεύσεις. Όλα αυτά μπορούν να κινητοποιηθούν περαιτέρω. Υπάρχουν και άλλα μέτρα, παραδείγματος χάρη της τυποποίησης ε, και αυτό έχει σχέση με τα μέτρα που προσφέρονται, ε, ο κανονισμός για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και μία σειρά και άλλων μέτρων, παραδείγματος χάρη κρατικές προμήθειες, ενωσιακά προγράμματα, πώς η διάσταση της ασφάλειας μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτά τα ενωσιακά προγράμματα. Ε, αυτό δεν είναι καινούριο, απλά ε, θέλουμε να το υπενθυμίσουμε, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ένα πιο ασφαλές δίκτυο ε, πέμπτης γενιάς τηλεπικοινωνιών. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς και τώρα θα ξεκινήσει η σειρά, η ε, ερωτήση από τους συντονιστές σε τρία λεπτά καθένας. από το ΕΛΚ, πρώτος, πρώτη μιλήτρια. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Όπως ε, ήδη αναφέρθηκε σήμερα, ε, η πέμπτη αυτή γενιά τηλεπικοινωνιών, δικτύων τηλεπικοινωνιών αλλάζει πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντική για την οικονομία και την κοινωνία. Ε, και θα είναι η ραχοκοκαλιά σε κρίσιμες ε, υπηρεσίες. Για να επιτύχουν όλα αυτά χρειαζόμαστε καθοδήγηση σε επίπεδο τεχνολογίες, χρειαζόμαστε ε, κανόνες, αυστηρούς κανόνες ε, που να είναι ηθικά βιώσιμοι και χρειαζόμαστε και εμπιστοσύνη. Και αυτή η ανακοίνωση είναι πολύ σημαντική για το θέμα της εμπιστοσύνης, για αυτό δηλαδή που συζητάμε. Έχουμε την αξιολόγηση κινδύνου και τέλος έχουμε πολύ σημαντικό ε, συστάσεις που απευθύνονται στα κράτη-μέλη. Η δική μου λοιπόν η ερώτηση είναι ε, πώς ακριβώς θα προχωρήσει η εφαρμογή όλων αυτών σε επίπεδο κρατών μελών. Δηλαδή τα κράτη-μέλη ε, θα αντιδράσουν γιατί υπάρχουν αρκετές διαφορές. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν Υπάρχει άραγε κάποια αρχή που να ελέγχει την εφαρμογή όλων αυτών των συστάσεων. Γιατί ε, πολύ ωραία όλα αυτά, ε, πολύ ωραία μελέτη, αλλά τι θα την κάνει κανείς αν δεν προβλέπεται και ακριβώς ε, πώς θα εφαρμοστούν οι συστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόγια για τους σοσιαλιστές. Όχι, εσείς παρακαλώ. καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη από τους προηγούμενους καλεσμένους, γιατί έφτασα αργά, έχει αλλάξει και η σειρά των σημείων της ημερήσιας διάταξη. Αυτό έκανα λάθος και μίλησα πριν για την τεχνολογία 5G. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, για την κατάσταση ασφάλειας ε, της πέμπτης γενιάς κινητών δικτύων τηλεπικοινωνιών. Τα κράτη-μέλη τώρα θα πρέπει να ανασκουμποθούν και να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν ε, τις μελλοντικές απειλές ε, που θα διαταράξουν ε, διάφορες πλευρές της καθημερινότητάς μας. Γιατί με τα αυτοματοποιημένα οχήματα σκεφτείτε τι κινδύνους θα αναλάβουμε αν δεν έχουμε μεριμνήσει για το θέμα της ασφάλειας. Νομίζω ότι η εργαλειοθήκη είναι κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και μπράβο σας. Ε, πάντως Είπατε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν να θεσπίσουν μέτρα και να ενισχύσουν ενδεχομένω τι αρμοδιότητε των ρυθμιστικών αρχών προκειμένου να αντιμετωπίσουν ε, αποτελεσματικά του κινδύνου. Ήδη στην ε, έκθεση του Οκτωβρίου είχατε τοπίσει κάποιου κινδύνου. Τώρα στα συμπεράσματα μα λέτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν κάποια μέτρα ασφάλεια. Ερωτώ λοιπόν το εξή. Ποιο είναι το επίπεδο τιμότητας στο οποίο βρισκόμαστε. Έχει προχωρήσει η θέσπιση των μέτρων, γιατί τον Απρίλιο, 30 Απριλίου, λίγη προθεσμία. Πώς θα εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της ενίας αγοράς, αν μια χώρα αποφασίσει να αποκλείσει μια επιχείρηση, ενώ άλλο κράτος δεν την αποκλείσει. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της παραβίασης της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών από πλευράς ε, εταιριών που ε, τα κράτη, οι εθνικές νομοθεσίες ε, υποχρεώνουν συνεργασία με τις επιχειρήσεις ό,τι αφορά την ανταλλαγή των δεδομένων για λόγους ασφάλειας και πώς εντάσσονται όλα αυτά στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι η Huawei θα μπορούσε και αυτή να συμμετάσχει στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που θα γίνουν για την εγκατάσταση του δικτύου 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι υπάρχουν αυστηρά κριτήρια και ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να απορρίψουν την υποψηφιότητα αυτή για ζητήματα ασφάλειας ή εξάρτησης. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε έναν κατάλληλο μηχανισμό αυτή τη στιγμή για να επαληθεύουμε τις κρατικές ενισχύσεις των τρίτων χωρών. Έτσι λοιπόν οι χώρες αυτές οι οποίες θέλουν να απομακρυνθούν από την Huawei ενδεχομένως να καθυστερήσουν πάρα πολύ στην εγκατάσταση του 5G όπως έχει συμβεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι μπορούν να προχωρήσουν σε εταιρική σχέση με την Ericsson, την Nokia και τις δύο εταιρείε. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που θα μπορούσαν να ελεγχθούν από τους Αμερικανούς είναι ότι η ευθύνη αυτή με την οποία επιβαρύνουμε τα κράτη-μέλη ενδεχομένως να δημιουργήσει μια γεωγραφική διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εγκατάσταση του 5G. Μήπως θα έπρεπε να ενισχύσουμε λίγο περισσότερο τις δικές μας ευρωπαϊκές εταιρείε, να μην περιμένουμε από τις Αμερικανικές να το κάνουν αυτό και μήπως η τελευταία ανάλυση ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να ευνοήσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείε που θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν τα δίκτυα των 5 5G. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των ε, Πρασίνων, ο κύριος Νινίστο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται, οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών όταν επενδύουν στο 5G ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ε, τιμές και ότι βασικά επιλέγουν ε, αυτόν που έχει να προσφέρει την πιο οικονομική προσφορά. Α μην ξεχνάμε όμω ότι είναι οι ευρωπαϊκέ εταιρείε αυτέ οι οποίε μπορούν να προσφέρουν τι πιο ασφαλεί λύσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή έχουμε μια τεχνολογική προσφορά η οποία είναι πιο ασφαλή, αλλά ενδεχομένω πιο δαπανηρή, πιο ακριβή. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δικιά τη επέμβαση να διορθώσει αυτή την ανισορροπία. Πρόεδρο, βλέπω ότι υπάρχει και εκπρόσωπο από την ομάδα ID. Θα σε το λόγο πριν από του πρασίνου. Ο κύριο Μποργία λοιπόν έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Κανένα πρόβλημα που ακούσαμε πρώτο τον προλαλήσαντα. Σε σχέση με την Huawei βλέπουμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά ότι έχουμε συγκεκριμένους κανόνες και οι κανόνες αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Και οι κανόνες είναι σαφέστατοι όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό και σε σχέση με την ακίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα που ουσιαστικά αναθέτει στα κράτη-μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένα μέτρα. Και πριν από μερικές μέρες η Huawei αποφάσισε να δημιουργήσει κάποια κέντρα παραγωγής στην Ευρώπη προκειμένου να καταφέρει να μετριάσει τον λεγόμενο ευρωπαϊκό σκεπτικισμό. Στο στάδιο λοιπόν αυτό, ένα στάδιο έντονης αμφισημίας, που φαίνεται και από τη στάση κάποιων κρατών μελών απέναντι στη Huawei. Νομίζω ότι αναδεικνύεται όλο και περισσότερο κάπως ο διστακτικός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών. Μήπως θα έπρεπε εδώ πέρα να καταφέρουμε να αντιταχθούμε κάπως την εμπορική στρατηγική πλέον που έχει αυτή η κινέζικη επιχείρηση και θεωρώ ότι είναι απόλυτα θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε με απόλυτη σαφήνεια για τους κινδύνους που ελοχεύουν στο πλαίσιο της εγκατάστασης του 5G από ξένες εταιρείες, εταιρείες τρίτων χωρών. Ωστόσο, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν θέλει να θίξει ευθέω την Huawei και θέλει να διατηρήσει απέναντί της μια διπλωματική, αν θέλετε, στάση, μήπως θα πρέπει να ανησυχούμε λίγο για την υγεία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πριν από λίγο καιρό, όταν είχαμε αυτή την έντονη αντιπαράθεση για τα δίκτυα 5G, υπήρχε μια επιχείρηση η οποία ξεκάθαρα είπε ότι αισθάνεται κάπως παραμελημένη Νομίζω λοιπόν ότι θα ήθελα εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει ένα κάποιο σχόλιο, καθότι η ανακοίνωσή σα αυτή υποτίθεται ότι θέλει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή έρευνα και τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Θα ήθελα να γνωρίσω τελικά αν οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με αυτά που έχουν να πούνε οι ίδιες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται, λαμβάνουν αυτή τη στιγμή περισσότερη υποστήριξη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν σε σχέση με το μηχανισμό ορίζοντας Ευρώπη 2020 σε σχέση με το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη θα μπορούσαμε να είχαμε μια πιο απτή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ως αναπληρωτή συντονιστής εξ ονόματος του ECR. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιο είναι το καθεστώς πραγματικά αυτής της εργαλειοθήκης για το μετριασμό των κινδύνων. Ξέρουμε ότι έχετε υποβάλει μια σύσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη είναι κάπως διχασμένα. Υπάρχουν χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία, η Εστονία που θα θέλανε πιο αυστηρούς ακόμα κανόνες. Αυτά τα οποία παρουσιάσατε είναι ελάχιστες απαιτήσει. Από την άλλη έχουμε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι άλλες χώρες οι οποίες θα προτιμούσαν πιο ευέλικτους ή λιγότερο αυστηρούς αν θέλετε κανόνες. Αυτή να θέλετε η πολιτική πτυχή. Υπάρχει κάποιος κοινό παρανομαστής σε αυτή την εργαλειοθήκη. Μιλάμε για κάποιες ελάχιστες απαιτήσει ασφάλειας τελικά. Και ένα δεύτερο ερώτημα όσον αφορά την λεγόμενη διατλαντική σχέση, τη σχέση που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο είπε ότι οι, Ευρω... οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα επέτρεπαν ποτέ την χρησιμοποίηση ενός ξένου δικτύου το οποίο δεν εμπιστευόμαστε, αναφερόμενο ουσιαστικά στο κινέζικο δίκτυο, στην κινέζικη τεχνολογία. Μπορεί η δική μας εργαλειοθήκη να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα ή μήπως αυτή η μηπω αυτη η διαφοροποιηση στη στάση τη εργαλειοθήκη που κρατούν τα κράτη-μέλη μπορεί να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά την εφαρμογή τη εργαλειοθήκη αυτή στην πράξη. Εξ ονόματο τη ΓκουΕ, τώρα υπάρχει κάποιο συνάδελφο που θα θέλει να πάρει το λόγο ω αντικαταστάτη του συντονιστή. Αν όχι, τότε α ακούσουμε του υπόλοιπου συναδέλφου. Ο κύριος Κρέμπλερ πρώτος. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την ΕΝΙΣΑ όσον αφορά την εργαλειοθήκη αυτή. Ξέρετε ότι η τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντική στον τομέα αυτό. Τα τελευταία 7 χρόνια έχω ασχοληθεί με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας και η συζήτηση γύρω από το 5G από τεχνικής πλευράς αφορά πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ασχολείται περισσότερο με την αρχιτεκτονική που, ασφαλείας που θα ακολουθηθεί. Ξέρετε ότι ε, πολύ συχνά και στο πλαίσιο του 4G το έχουμε πει αυτό, ότι υπάρχει αν θέλετε ένας διακόπτης ενεργοποίησης του συστήματος. Αν λοιπόν υπάρχει μία εταιρεία που χειρίζεται το σύστημα αυτό, ενδεχομένως να είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση του 5G παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε εμείς ότι ε, οι εταιρείε αυτές δεν θα λειτουργήσουν οριζοντίως και εντελώ εικονικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε από το 5G οποιαδήποτε χώρα η οποία θα μπορούσε να στραφεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κυβερνοχώρο. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη διάκριση ανάμεσα στο κεντρικό σύστημα και στο το σύστημα των παρυφών, του δικτύου παρυφών. Νομίζω ότι εδώ πέρα πάλι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να αποκλείσει εταιρείε όπω η Highway. Αν ενεργοποιηθεί μια τέτοια εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε προφανώ, έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε. Κυρία Τόια, τώρα έχει το λόγο. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα στον, ε, ε, ε στον ε, Υποθέτω ότι αυτή η νέα τεχνολογία, μάλλον να σας πω ότι ήμουν εισηγήτρια, εισηγήτρια για αυτή την τεχνολογία ε, γιατί χωρίς αυτή τη τεχνολογία δεν θα υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε χρήση αυτής, αυτού του δικτύου. Ε, τώρα όμως πρέπει να σας πω ότι έχω κάποιες αμφιβολίες. Το πρώτο είναι, βεβαίως, ε, βλέποντας το τι μας είπατε, ε, θέλω να ρωτήσω το εξή. Κάναμε όλες τις επαληθεύσεις για την ασφάλεια από πλευράς υγείας, αν θέλετε, της τεχνολογίας. Αυτή είναι μια ερώτηση που την έκανα και προς την Κομισιόν. Και αυτό το λέω όχι για να τον μπλοκάρουμε το 5G, αλλά για να ξέρουμε όλοι τι συνεπάγεται. Γιατί υπάρχουν όλες αυτές τις δυνατότητες ε, πρόσβασης, η πλήρης κάλυψη. Υπάρχει λοιπόν μια διάχυση που θα έλεγα πολύ σημαντική διάχυση ηλεκτρομαγνητική. Εγώ απλά θέλω να το ρωτήσω και η δεύτερη ερώτηση αφορά το θέμα του χώρου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Επιτροπή αυτή ασχολούμεθα με το χώρο, είναι πολύ σημαντικό. Ε, το 5G ε, νομίζω ότι χρησιμοποιεί περίπου την ίδια χωρητικότητα όπως το πρόγραμμα Γαλιλαίος και Κοπέρνικους. Μήπως λοιπόν λοιπόν θα υπάρχουν ε, προβλήματα επικοινωνίας με αυτά τα δύο διφορικά συστήματα. Το έχετε αυτό ελέγξει ή όχι. Και τέλος, μια πολιτική οικονομική ε, ερώτηση, δηλαδή ε, είχαμε δει ότι υπάρχει μία πίεση από τους φορείς εκμετάλλευσης, ε, κυρίως από αυτούς που ενδιαφέρονται. Ε, αν το λιγάκι την εισήγησή σας, ε, γίνεται λόγος για το ότι αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη έχουν διαθέσει ένα μεγάλο ποσοστό περίπου το 16% ε, και θέλω να ρωτήσω υπάρχει κάποια επιφύλαξη ε, από τις φορείς εκμετάλλευσης ε, να μην θέλουν να δαπανίσουν όλο αυτό το χώρο και να περιμένουν λιγάκι τι θα γίνει με τους δημόσιους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν. Σας ευχαριστώ. Χαιρετίζω και εγώ την εργαλειοθήκη για το μετριασμό των κινδύνων στην τεχνολογία πέμπτης γενιάς κινητών δικτύων. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ενσαρκώνει τον ευρωπαϊκό τρίτο τρόπο. Γίναμε μάρτυρες μιας ανοιχτής αντιπαράθεσης μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς στην Ευρώπη. Το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θέτησαν μονομερείς αποφάσεις για την πρόσβαση ξένων προμηθευτών τεχνολογίας πέμπτης γενιάς. Και μια και η εργαλειοθήκη περιέχει συστάσεις και είναι ε, προαιρετικού χαρακτήρα. Πώς θα αποφύγουμε τον πιθανό κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς με αυτές τις μεμονωμένες και μονομέρειες αποφάσεις των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάπτυξη της τεχνολογίας πέμπτης γενιάς και τη χρήση της εργαλειοθήκης, στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι θα λάβει υπόψη και τις επιπτώσεις στην υγεία. Φαίνεται όμως ότι μέχρι στιγμής ε, παραβλέπεται αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία. Δεν έχουμε πραγματοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση καν μία μελέτη αντικτύπου της τεχνολογίας αυτής στην υγεία του ε, ανθρώπου αλλά και στο περιβάλλον. Ενώ κάποιες χώρες όπως το Βέλγιο για παράδειγμα ε, έχουν επιβάλλει δικαιοστάσιο στις τεχνολογίες πέμπτης γενιάς εν ώψη αναμονής ε, μελετών αντικτύπου για την τεχνολογία 5G. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς στην Ευρώπη. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε ευρηματικές και καινοτόμες τεχνολογικές ε, λύσεις και το χάσμα με τους υπόλοιπους ε, διεθνείς παράγοντες θα αυξάνεται. Θα πρέπει όμως όλοι οι Ευρωπαίοι να αποφεληθούν από την πέμπτη γενιά και να έχουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη και γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη της πέμπτης γενιάς των κινητών δικτύων τηλεπικοινωνιών. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει μια κοινή προσέγγιση πραγματικά πανευρωπαϊκή, γιατί τα κράτη-μέλη ε, αναλαμβάνουν ε, μονομερείς αποφάσεις και τέτοια μεμονωμένη πολιτική των κρατών μελών ε, υπονομεύει την ανάγκη κοινή προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Σοχίνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστέρησε η πτήση μου και δεν πρόλαβα να ακούσω την αρχική παρουσίαση. Θα ήθελα όμως ε, να σας παρουσιάσω μια σκέψη μου. Εξέτασα τα έγγραφα και φαίνεται ότι γίνεται μια σημαντική συντονισμένη προσπάθεια ώστε η νέα αυτή τεχνολογική φάση να έχει και μια κοινωνική διάσταση και η ασφάλεια να συνδυαστεί με ηθικές και δοντολογικές αξίες και την εξυπηρέτηση των Ευρωπαίων πολιτών για να δει ο Ευρωπαίος πολίτης, πού έγκυται η διαφορά του ευρωπαϊκού μοντέλου σε σχέση με τα άλλα. Και μάλιστα ήμουν και εισηγητής μιας έκθεσης πρωτοβουλίας, της πρωτοβουλίας Wi-Fi for EU. Και ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιλωτική εφαρμογή του Wi-Fi for You e που εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Και προβλέποντα κάποιες φάσεις του πιλωτικού προγράμματος, όχι μόνο για τις κεραίες, αλλά και μετά για νέο σύστημα για όλη την Ευρώπη. Και έχουμε μεγάλη ευκαιρία να έχουμε ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα και για ε, το 5G που θα δίνει την ταυτότητα της Ευρώπης. Γιατί το Wi-Fi for You έγινε σημείο αναφοράς και θα συνεχιστεί. Αλλά στα έγγραφά σας δεν βλέπω καμία ε, μνήα αυτού του προγράμματος. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που ήταν επιτυχημένο και να γίνει ένα σημείο αναφοράς και για την τεχνολογία 5G που θα πρέπει να βρεθεί στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τους συναδέλφους και θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Γκονσάλες Ποντέρο, Σάντσο Ποντέρο, για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι. Τις κατέγραψα προσεκτικά και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις απορίες σας. Η κυρία Καρβάλιο έθεσε ερωτήσεις ε, για το βαθμό εφαρμογής των μέτρων της εργαλειοθήκης. Η εργαλειοθήκη, επαναλαμβάνω, αποτελεί τον καρπό συνένεσης. Είναι ένα έργο στο οποίο συμφώνησαν τα κρατημέλη και μόλις εγκρίθηκε. Βέβαια, από πολιτικής άποψης ε, είχαμε ταχύς ρυθμός ε, πρόοδου. Γιατί το να καταλήξουν τα κράτη-μέλη, ο ΕΝΗΣΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια κοινή προσέγγιση και κοινά μέτρα και κοινή μεθοδολογία αυτό από ευρωπαϊκή άποψη ήταν αστρονομική ταχύτητα, σχεδόν ταχύτητα διαδικτύου. Και μάλιστα στην ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είστε στα κράτη-μέλη μέχρι τις 30 Απριλίου να λάβουν, να υιοθετήσουν κάποια μέτρα. 30 Απριλίου είναι σχετικά σύντομη η προθεσμία. Και κανένα κράτο μέλο δεν διαμαρτυρήθηκε ότι είναι πολύ σύντομη αυτή η προθεσμία. Φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει τα κρατημέλη να επιταχύνουν του ρυθμού. Και ένα από τα μέτρα που αναφέρουμε στην ανακοίνωση είναι να συστήσουμε μία ομάδα που είχε γίνει ad hoc για το συγκεκριμένο θέμα να μονιμοποιηθεί για τη συνεργασία στην ασφάλεια των δικτύων 5G. Αποφασίσαμε να μονιμοποιήσουμε αυτή την ομάδα εργασία και. Ήδη την Πέμπτη θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε συνεχίζουμε με αμύωτο ρυθμό. Πολλοί ευρωβουλευτές έθεσαν την ίδια ερώτηση για την παρακολούθηση, το monitoring και τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι φυσικά υπάρχει εσωτερική αγορά Φυσικά και προέχει η συνοχή και η ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς, αλλά μιλούμε και για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και κάποιες πτυχές της εθνικής ασφάλειας ε, ε, είναι εθνική αρμοδιότητα. Και εκεί υπάρχουν διαφορές. Αλλά τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια κοινή προσέγγιση που ναι μεν δεν είναι νομικά δεσμευτική, αλλά πολιτικά είναι δεσμευτική. Γιατί τα κράτη-μέλη συναποφάσισαν ε, προσυπέγραψαν αυτό το έγγραφο της εργαλειοθήκης και τη μεθοδολογία. Και φυσικά ένα κράτος μπορεί να συμφωνήσει σε ένα έγγραφο και να μην το εφαρμόσει, αλλά θα πρέπει να αιτιολογήσει τη θέση του, αν το κάνει. Και σίγουρα η παρακολούθηση είναι σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας, σημαντικό τμήμα της διαδικασίας. Και δεν είμαστε εδώ στη λογική ότι η Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την υιοθετούν και ελέγχουμε την ε, εφαρμογή. Η παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική γιατί τα κράτη-μέλη θέλουν να συνεργαστούν και να συγκρίνουν τις προσπάθειές τους. Άλλα είναι πιο προηγμένα και άλλα όχι τόσο. Γι' αυτό και η παρακολούθηση αποτελεί κεντρικό σημείο της διαδικασίας. Τώρα, το επίπεδο ετοιμότητας και εκεί υπάρχουν διαφορές. Πόσο προετοιμασμένα είναι τα κράτη-μέλη ε, ένα συγκεκριμένο κράτος που είναι πια πρώην κράτος έχει εδώ και χρόνια εφαρμόσει ένα σύστημα για την παρακολούθηση της ασφάλειας, ιδιαίτερα για τις αλλοδαπές εταιρείε. Οπότε είχε πολλές εμπειρίες. Σε άλλα κράτη δεν υπάρχει τέτοια εμπειρία. Εξού και το ενδιαφέρον της σύγκρισης των προσεγγίσεων των εθνικών. Και υπάρχουν διαφορές, όντως υπάρχουν διαφορές, αλλά το όλο σκεπτικό της προσέγγισης είναι, είναι κοινή αλλά να μπορεί να προσαρμόζεται στις διαφορές των κρατών μελών και σε επίπεδο προθεσμιών και χρονοδιαγράμματος. Σε μερικές περιπτώσεις τα μέτρα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια εφόσον καθυστερήσουν κάπως οι πολιτικές αποφάσεις. Επίσης, πώς θα προστατευτούμε από παραβιάσεις της εμπιστευτικότητας. Αυτό το αναφέραμε και στην αξιολόγηση κινδύνου του Οκτωβρίου. Η πιθανή παρέμβαση παραγόντων από τρίτες χώρες είναι συγκεκριμένος κίνδυνος και το επισημάναμε. Και η πιστοποίηση αναφέρεται σε διάφορα σημεία της εργαλειοθήκης και είναι ένα από τα μέτρα που μπορεί να εθετηθεί. Η πιστοποίηση των τεχνολογιών 5G και των διαφόρων πτυχών τους. Ε, είναι ένα θέμα που έχουμε επισημάνει. Και τρεις ερωτήσεις αφορούσαν και πάλι τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Όντως υπάρχουν διαφορές, αλλά επαναλαμβάνω, το όλο σκεπτικό ήταν να έχουμε μια προσέγγιση βάσει συνένεση, συμφωνίας και η εφαρμογή να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες. Υποστήριξη των Ευρωπαίων προμηθευτών η ευρωπαϊκή προτίμηση, η προτίμηση στους Ευρωπαίους προμηθευτές. Φυσικά η γραμμή εδώ είναι ξεκάθαρη. Η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή αγορά, οπότε οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Ε, και τηρώντας φυσικά τους κανόνες, αυτό είναι απαράβατη αρχή. Και αυτό που αναφέρουμε στην ανακοίνωση, το θέμα της ασφάλειας ε, είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στους μελλοντικού μας διαγωνισμούς. Αυτό θα το λάβουμε υπόψη. Οπότε δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται κάποια προγράμματα. Και ήδη σε πολλά προγράμματα χρηματοδότησης υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις και διατάξεις. Ίσως θα πρέπει να περιλάβουμε και νέες διατάξεις ενδεχομένω, ειδικά για το θέμα της ασφάλειας της τεχνολογίας 5G. Τώρα, ευρωπαϊκές εταιρείε ενδιαφέρονται περισσότερο για την τιμή και όχι τόσο για την ασφάλεια. Σίγουρα, αν παραμελήσουμε την ασφάλεια, θα μας στοιχήσει πολύ ακριβά στο μέλλον. Οπότε υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη ω προς αυτό το σημείο. Η ασφάλεια δεν είναι, η ασφάλεια δεν είναι κάτι αφηρημένο. Και πραγματικά η, αλλαγή στην πολιτική συζήτηση δείχνει ότι η ασφάλεια δεν είναι πια ζήτημα τεχνικών τμήματων και μονάδων μόνο, αλλά είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλες τις εταιρείε και σίγουρα και οι εθνικές αρχές εγκύπτουν με ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της ασφάλειας. Αναφέρθηκε μία συγκεκριμένη εταιρεία, ε, όχι εταιρεία, του εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίζει περισσότερο τους Ευρωπαίους προμηθευτές και αν υπάρχει βούληση για κάτι τέτοιο. Σας είπα και προηγουμένως, στην ανακοίνωσή μας αναφέρονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης της καινοτομίας. Και μέσω αυτών των προγραμμάτων λαμβάνουμε υπόψη και θέματα ασφάλειας. Κάποιος ευρωβουλευτής είπε ότι δεν έχουμε κάποιο μηχανισμό για να καταπολεμούμε επενδύσεις ξένων ε, επιδοτήσεις ξένων κυβερνήσεων. Κι όμως έχουμε, γιατί μιλούμε για αποφυγή της τρέβλης εσωτερικής αγοράς λόγω επιδοτούμενων ε, εισαγωγών ή εισαγωγών σε τιμές dumping. Υπάρχει μηχανισμός που μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δημιουργείται στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς λόγω τέτοιων ξένων επιδοτήσεων. Και η εργαλειοθήκη δεν είναι πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επαναλαμβάνω, είναι καρπός ε, της ομάδας συνεργασίας ε, της Οδηγίας ΝΙΣ για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Ε, στην ομάδα αυτή προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Κροατικής Προεδρίας και συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΕΝΙΣΑ και τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό σε αυτή την ομάδα εργασίας. Και η εργαλειοθήκη δεν είναι νομικά δεσμευτικό κείμενο, αλλά πολιτικά δεσμευτικό. Και μερικές φορές η πολιτική δέσμευση είναι εξίσου σημαντική, ίσως και σημαντικότερη και από την νομική δεσμευτικότητα ή ισχύ ενός εγγράφου. Τώρα, κάποιο μίλησε για τι διατλαντικέ σχέσει. Αναφέρθηκε και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, και τι δηλώσει του. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία στην Ευρώπη όταν αντιδράσαμε ε, στις πιέσεις ή αιτήσει ε, κάποιων εταίρων μας από την Κίνα, από την ΗΠΑ. Και είπαμε κάτι πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι τα κράτη-μέλη θα συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνουμε μία ανάλυση βάση κινδύνου. Και ήταν μια διαδικασία που έγινε γρήγορα, αλλά χωρίς υπερβολική βιασύνη. Και μάλιστα και ο Μαρκ Πομπέο χαιρέτησε την εργαλειοθήκη και τα ενδιαφερόμενα μέρη το ίδιο. Το θέμα βέβαια είναι η εφαρμογή της εργαλειοθήκης. Όλοι μέχρι στιγμή εργαστήκαμε πολύ καλά, το επόμενο βήμα θα είναι η εκτέλεση των μέτρων αυτών, των συστάσεων. Τέθη ένα ερώτημα ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στον πυρήνα και στις παρυφές. Ε, ίσως λοιπόν ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε να αποκλείσουμε ε, παρόχους υψηλού κινδύνου. Και αυτό ήταν στον πυρήνα της ανάλυσης. Δηλαδή ποια είναι τα ευαίσθητα εκείνα θέματα, πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τους κινδύνους, η προσέγγιση ε, αφορά κάποιες ε, λεπτομέρειες και όσον αφορά αυτές τις διαφορετικές θέσεις, πράγματι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Σε τελική ανάλυση αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ένας κατάλογος, μια ανάλυση και με βάση αυτήν την ανάλυση να εφαρμοστούν τα μέτρα. Υπάρχουν και κάποιες ε, ερωτήσεις, κυρίως αυτές που έθεσε η κυρία Τρόγια, που αφορούν σε θέματα τα οποία δεν καλύπτονται στην ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αφορά την ασφάλεια. Τίθεται το θέμα της υγείας ε, των ανθρώπων. Πράγματι γίνεται δουλειά επ' αυτού. Υπάρχουν ε, ε, κάποιες συστάσεις που ανάγονται στο 99 και συνεχίζεται η δουλειά πάνω σε αυτές τις συστάσεις. Προσπαθούμε να τις εξετάσουμε. Έχουμε ακούσει διάφορες απόψεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το θέμα. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται το διάλογο με τον ε, ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κυρίως με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος για αυτά. Όσον αφορά τα δίκτυα, ε, το 60% ε, είναι πιλωτικά δίκτυα και εμείς πιστεύουμε ότι ο ρυθμός εφαρμογής ε, των αποφάσεων για το σύστημα 5G πάει πάρα πολύ καλά, αλλά διάφορα κράτη-μέλη περιμένουν το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς για να μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις τους. Σχετικά με, την, ε, με τις παρεμβολές με το πρόγραμμα Κοπέρνικος και Γαλαίος, φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω τίποτα από αυτού. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα είναι εκείνε ε, που ε, καταδεικνύουν ότι τα κράτη-μέλη ακολουθούν τελείω διαφορετικό δρόμο. Υπάρχουν διάφορε ευαισθησίε, αλλά και όλοι αυτοί έχουν αποφασίσει να στηρίξουν αυτό το έγγραφο. Και πάλι για το θέμα τη υγεία, μήπω έχει αγνοηθεί το θέμα τη υγεία. Σα απάντησα ότι το θέμα εξετάζεται και ίσω πρέπει να υπάρξει εμβάθυνση στο θέμα αυτό. Κοινή προσέγγιση, νομίζω ότι υπήρξε απάντηση σε αυτό. Και τέλος ε, το Wi-Fi for you, ε, ποια είναι η αναλογική σχέση με αυτό το σύστημα και ποια είναι τα μαθήματα που προκύπτουν από αυτό όταν μιλάμε για, μιλάμε για διαφορετική τεχνολογία, τουλάχιστον όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ε, αναλογία ίσως να υπάρχει στην προσέγγιση ως προς την υποστήριξη που μπορεί να προσφερθεί στην ε, Ευρώπη. Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξαστεί. Νομίζω ότι λίγο πολύ κάλυψα όλες τις ε, ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε άλλα 10 λεπτά. Αν ε, υπάρχουν κάποιες επίγουσες ερωτήσεις, παρακαλώ μην διστάστε να τις ε, θέσετε. Αν όχι, τότε ολοκληρώθηκε αυτό το σκέλος της, ε, των εργασιών μας. So now we are going to the next item, uh, item 5, it is a report from Commission and the European Parliament. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που αφορά τα θέματα της ε, περιαγωγής. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Βέζα Τεράβα, ο οποίος ε, είναι εκτελή χρέη διευθυντού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να σας υπενθυμίσω ότι ε, ο κανονισμός για την περιεγωγή υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και οι νέοι κανόνες ε, ε, υποβλήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου του 2019. Είχαμε και μία ενδιάμεση εξέταση του θέματος της λειτουργίας της αγοράς περιαγωγής. Για το θέμα αυτό έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και τα ήθελα και για άλλη μια φορά να σας καλέσω να δείξετε το ενδιαφέρον σας λαμβάνοντας το λόγο. Και τώρα λοιπόν ξεκινάμε με την παρουσίαση. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, ενημερώσω σχετικά με τα θέματα περιαγωγής, ε, κυρίως όσον αφορά την έκθεση που υιοθέτησε η Επιτροπή τέλη Νοεμβρίου. Και η έκθεση αυτή αφορά στην εφαρμογή του κανονισμού για την ε, περιαγωγή, ε, κυρίως για την περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού, η οποία έχει αφήσει εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2017. Όσον αφορά την έκθεση που υιοθετήσαμε τον Νοέμβρη, θέλω να σας πω ότι εξετάσαμε τα δεδομένα, είδαμε τις εκθέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής και επίσης διεξαγάγαμε και μία μελέτη. Με λίγα λόγια λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, με λίγα λόγια και πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε αυτά που βλέπεις στη διαφάνεια και μετά θα μπω σε λεπτομέρειες. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το καθεστώς της περιεγωγής με χρέος εσωτερικού, αυτό ήταν πετυχημένο, μεγάλη επιτυχία για τους ε, τελικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τις ε, μικρές ε, επιχειρήσεις όπως έδειξε και η έκθεση του Κοινοβουλίου οι φορείς εκμετάλλευσης είναι ευχαριστημένοι, επέδειξαν πνεύμα εργασία, συμμορφώθηκαν με τους κανόνες και τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή των ε, κανόνων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επέλυσαν τα θέματα ε, ταχύτατα. Ως εκ τούτου το τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό. Αργότερα θα αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως η αγορά χονδρικής ε, είναι πολύ σημαντική για να μπορεί να λειτουργεί και η αγορά λιανικής. Η αγορά χονδρικής πρώτα απ' όλα κατέδειξε ότι τα τέλη περιαγωγής χονδρικής μειώθηκαν μειώθηκαν σημαντικά. Μειώθηκαν βέβαια σημαντικά ε, γιατί ε, επιβλήθηκαν κανόνες ε, στους φορείς εκμετάλλευσης. Όμως τελικά τα τέλη που καταβάλουν οι πάροχοι για τις υπηρεσίε περιεγωγής, αυτά τα τέλη είναι χαμηλότερα από αυτά που είχαν προβλεφθεί. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι πάροχοι μπορούσαν να καλύψουν τις δαπάνες τους. Τίθε το ερώτημα. Αυτοί οι πάροχοι που δεν έχουν το δικό τους το δίκτυο, αυτοί πώς μπορούν ε, να αντιμετωπίσουν το νέο καθεστώς. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών μπόρεσαν να διατηρήσουν το κομμάτι τους, το μερίδιο τους στην αγορά. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ε, υπάρχει μεγάλο βάρος ε, από την εφαρμογή των κανόνων. Επίσης, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι πάροχη ε, πάροχοι των ε, κινητών υπηρεσιών μπορούν να τα καταφέρουν. Ε, πάρα πολλοί από του φορεί εκμετάλλευση δικτύου κινητών επικοινωνιών έχουν παραμείνει μέσα στα ανώτατα όρια. Άρα δηλαδή οι μελέτε δείχνουν ότι τα αποτελέσματα είναι καλά, καλά γιατί είναι και σωστοί οι κανόνες. Ε, ο Ε, οδήγησε στο ότι η περιαγωγή ήταν επιτυχημένη. Αλλά αν δεν υπήρχαν οι κανόνες και οι κανονισμοί δεν θα υπήρχε αυτή η επιτυχία. Να μπω σε λεπτομέρειες. Τώρα όσον αφορά την αγορά λιανικής, αυτό που είδαμε μετά την εισαγωγή του συστήματος περιαγωγή με χρέο ιστορικού, μειώθηκαν σημαντικά τα τέλη, ε, τριπλάσια η ε, μείωση ε, στα φωνητικά μηνύματα, αλλά εξίσου ε, σημαντική μείωση και στην διακίνηση των δεδομένων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι αυτό το σύστημα της περιεγωγής με χρέο εσωτερικού, αυτό ήταν ένα ευπρόσδεκτο σύστημα από τους τελικούς χρήστες, οι οποίοι πλέον δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες παραγωγής όταν ταξιδεύουν σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστημένοι καταναλωτές, αυτό το έδειξε και το βαρόμετρο, το Ευρωπαϊκό μετρό, Βαρόμετρο, ε, έγιναν οι σχετικές έρευνες και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι τελικά υπήρξαν κέρδη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατόπιν, όταν διαπραγματευθήκαμε τους ε, κανόνες, γίνονται συζητήσεις για το κατά πόσον ο κανονισμός για την ε, επιβολή των ε, τελών περιεγωγής να είναι όπως αυτά του εσωτερικού, κατά αυτό θα οδηγούσε ενδεχομένως σε αύξηση άλλων τελών, κυρίως αυτών για τις τρίτες χώρες ή ε, για στα τέλη ε, εσωτερικού. Βλέπουμε όμως ότι και αυτός ο κίνδυνος ήταν ε, υπερτιμημένος. Βλέπουμε να υπάρχει πτωτική τάση στις εσωτερικές τιμές και επίσης τα τέλη περιεγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται και αυτά σε πτωτική τροχιά. Στον κανονισμό για την περιαγωγή έχουμε δικλείδες ασφαλείας για τους παρόχους για να μπορούν και αυτοί να διαφυλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Έχουμε τη νέα πολιτική και από την άλλη έχουμε και νέες δυνατότητες επιλογής. Έτσι λοιπόν οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν τη δυνατότητα να αποκλίνουν ε, από την περιεγωγή με χρέο εσωτερικού στο βαθμό που αυτή η περιαγωγή πλήττει την κερδοφορία τους. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα αυτή, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση κάποιων πολιτικών αποτυχίας, 95% για τους MNOs και 78% όσον αφορά τους MVNOs, που έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την πολιτική της εύλογης χρήσης. Πρέπει όμως να παρατηρήσουμε και το ακόλουθο ότι ε, η ε, κίνηση περιαγωγής αυτή τη στιγμή συνδυάζεται με την πολιτική εύλογης χρήσης εφαρμόζεται σε ένα 6% του, ε, της κίνησης φωνητικών δεδομένων και 4% για τα δεδομένα. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ένα 95% όλη της κυκλοφορία δεδομένων προσφέρεται τελικά σε εγχώριε τιμέ. Από πλευράς λοιπόν τελικού χρήστη είχαμε ελάχιστε ε, μόνο περιπτώσεις ε, όπου ε, η ποσότητα αυτή κυκλοφορίας πραγματικά εμπίπτει στην πολιτική ευλογής χρήση, στην παρέκκληση βιωσιμότητος. Και εδώ είχαμε μόνο 1,5% όσον αφορά την κυκλοφορία δεδομένων και περίπου 3% όσον αφορά την κίνηση φωντικών δεδομένων. Δηλαδή, μόνο στι περιπτώσει αυτέ χρησιμοποιήθηκε η παρέκκληση βιωσιμότητο και είχαμε επιπλέον επιβάρυνση. Τώρα, όσον αφορά ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίω αν οι υπηρεσίε αυτέ έχουν κάνει δεδομένα. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε θεμελιώδη ζητήματα όπως ε, το βριζονικό δίκτυο ή ταχύτητα. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό για την παροχή της υπηρεσίας της ίδιας ακόμα και αν δεν πληρώνει κανείς επιπλέον τέλη. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε εδώ πέρα είναι ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, 14 σε σύνολο 30 εθνικών ρυθμιστικών αρχών έχουν καταγράψει καταγγελίες των καταναλωτών ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γνωμοδότης της Μπέρεκ αναφέρεται σε μια απουσία διαφάνειας όσον αφορά τις εκθέσεις για την ποιότητα των δεδομένων. Και πάλι όμως εδώ πέρα η παρατήρηση αυτή που έχει να κάνει με την ταχύτητα των δεδομένων, η οποία ενδεχομένω να είναι χαμηλότερη όταν είναι κανεί σε συνθήκε περιαγωγή, είναι μια παρατήρηση που έχει κάνει το Μπέρεκ και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ακόμα περισσότερο. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια δεδομένα όσον αφορά τα ανώτατα όρια τιμών χονδρική περιαγωγή 4,5 ευρώ ανά γίγαμπιτ μειώνονται σε 3 ευρώ αργότερα και βλέπουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση 2,5 ευρώ για το 2022. Ενδεχομένω η γραφική αυτή παράσταση είναι κάπως περίπλοκη. Έχουμε εδώ πέρα δεδομένα από το 2019 όταν είχαμε ένα χάσμα 6% 6 ευρώ μάλλον γιγαμπάιτ. Βλέπετε εδώ πέρα ότι και πάλι οι τιμές οι οποίες προτείνονται από τα κράτη-μέλη είναι χαμηλότερες από τις ανώτες τιμές χονδρικής περιαγωγής. Οι πραγματικά καταβληθήσεις, δηλαδή τιμές χονδρικής περιαγωγής, είναι χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες ανώτες τιμές. Βλέπετε εδώ πέρα, με διαφορετικό χρώμα, τα δεδομένα για τους MVNOs, MVNOs με πορτοκαλί και με μπλε MNOs. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν κάποιες κουκίδες οι οποίες βρίσκονται κάτω από τη διαχωριστική αυτή γραμμή. Υπήρχαν δηλαδή και MNOs e οι οποίοι κατάφεραν να παρέχουν τιμέ, να προτείνουν τιμέ οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις ανώτατες τιμές χονδρικής περιεγωγής. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία των MVNOs στην αγορά. Βλέπετε εδώ πέρα ότι οι MVNOs, ε, οι φορείς εκμετάλλευση εικονικού δικτύου κινητών επικοινωνιών, δεν έχουν χάσει τελικά τα συνολικά μερίδια αγοράς που είχαν, τα οποία έχουν παραμείνουν πάνω κάτω τα ίδια και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ε, υπάρχουν και κάποιοι MVNOs που κατάφεραν τελικά να αυξήσουν ε, το μερίδιο αγοράς τους. Το βλέπετε αυτό στις κουκίδες που είναι αριστερά της διαχωριστικής γραμμής. Και μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τόσο όσον αφορά την περιεγωγή λιανικής και όσον αφορά την ε, περιεγωγή χοντρικής, οι επιπτώσεις ήταν θετικές για του MVNO που κατάφεραν, όπω σα είπα, να διατηρήσουν το μερίδιο αγορά του. Έχετε εδώ μια πολύχρωμη γραφική παράσταση, η οποία καταδεικνύει την κατάσταση σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν γέννη, από τη γραφική αυτή παράσταση μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα το οποίο σα παρέθεσα πριν από λίγο, ότι οι πραγματικέ τιμέ χονδρική παρουσιάζουν μείωση και ότι ε, το γενικότερο κόστος παρουσιάζει και αυτό καθοδική τάση. Ας περάσουμε τώρα σε κάποια τελικά συμπεράσματα. Όπως είπα στην αρχή της παρουσίασής μου, η επισκόπηση, δική μας η αξιολόγηση και η αξιολόγηση που έκανε και η Μπέρεκ, ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τίποτα δεν έχει τροποποιηθεί πέρα από τις ρυθμισμένες προϋποθέσεις. Έχουμε κρατήσει την δυναμική ανταγωνισμού Πρέπει εδώ πέρα όμως να ρωτηθούμε τι θα γίνει όταν λήξει το 2022 ο κανονισμός. Αν θα πρέπει να υπάρξει κάποια άλλη ρυθμιστική, ε, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα αντικαταστήσει τον κανονισμό αυτό για να αποφύγουμε μια αύξηση των τιμών. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανεί πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Πάντως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα αναθεωρήσουμε τον εν λόγω κανονισμό. Επίση, Είδαμε τα όσα έχουν συμβεί και όσα συμβαίνουν επί του παρόντος στην εν λόγω αγορά περιαγωγής. Έχουμε τη χρησιμοποίηση όλο και περισσότερο του διαδικτύου των πραγμάτων, όλο και περισσότερες διαδικτυακές ηλεκτρονικές εφαρμογές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μόνιμη πλέον περιαγωγή. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, όλο και περισσότερο φορείς που χρησιμοποιούν την περιαγωγή σε μόνιμη βάση, κάτι το οποίο δεν καλύπτεται από τον κανονισμό, ο οποίος κανονισμός αναφέρεται μόνο στις, στα προσωρινά ταξίδια, στην προσωρινή διαμονή σε μια άλλη χώρα και επομένω καλύπτει την ε, προσωρινή περιαγωγή και όχι τη μόνιμη περιαγωγή και επίσης ε, οι συμβάσεις ε, μεταξύ των διαφορετικών φορέων εκμετάλλευσης βασίζονται σε καθαρά εμπορικού όρους αυτή τη στιγμή. Έπειτα έχουμε και την ρήτρα λήξη ισχύω ε, όσον αφορά τον κανονισμό περιαγωγής. Θα τέλη Ιουνίου του 2022 λύγει ο κανονισμός αυτός, που ήδη από τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Θα πρέπει να καταλήξουμε πρώτα σε μια τοποθέτηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενέστε δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον και ενδεχομένω να έχετε δει ότι στο πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη για φέτο, για το 2020, προβλέπεται η αναθεώρηση του κανονισμού περιαγωγή μέχρι τα τέλη του τρέχοντο έτου. Ξεκινάμε λοιπόν την όλη διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης και μέσα στους επόμενους μήνες και με τη μελέτη αντικτύπου που καθώ επίση και με τη δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσει πολύ γρήγορα, θα είμαστε σε θέση στα τέλη του έτους να καταλήξουμε σε κάποια εσωτερικά συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουμε με τον κανονισμό για την περιαγωγή από τη στιγμή που θα λήξει. Και βέβαια, αν καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση, θα πρέπει να προβλέψουμε και τον το χρόνο προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορέσουν και αυτά να αντιδράσουν σε σχέση με τη δική μας πρόταση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Βέσα Ταρόβα για την παρουσίασή σας. Περνάμε σε ερωτήσεις των συντονιστών από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κυρία Μέιντελ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Χαίρομαι που συζητάμε κάτι που μας απασχόλησε στο παρελθόν και το επιδιώξαμε και μας χαροποιεί το ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που αναφέρατε κι εσείς. Τον Ιούνιο του 2017, με την κατάργηση των τελών περιαγωγής, είχαμε δωδεκαπλάσια αύξηση του όγκου των κινητών δεδομένων στην Ευρώπη εντυπωσιακή αύξηση και ο ρυθμός και των τηλεφωνημάτων διπλασιάστηκε. Οπότε είναι σαφές ότι η νομοθεσία αυτή ήταν απαραίτητη και γι' αυτό και την προωθήσαμε τόσο πολύ. Και τα τελευταία δύο χρόνια έχουν φανεί τα θετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Και καλό θα είναι τέτοιου είδους ε, επιτεύγματα να κοινοποιούνται και προς τα έξω, να μην μένουν εντός των τυχών του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Είναι ένα από το παράδειγμα μιας κοινοτική ρύθμισης που ωφελεί τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, ο κανονισμός δείχνει και την τεράστια πρόοδο που έχουν κάνει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα προκειμένου να άρουν κάποια εμπόδια και φραγμούς της εσωτερικής αγοράς και να την υλοποιήσουν στο έπακρο. Και είναι επίσης το είδος της νομοθεσίας που ενισχύει και την ανταγωνιστικότητα ταυτόχρονα. Και εξασφαλίζει καλύτερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο παγκόσμιο προσκήνιο. Κάτι που βοηθά τις ευρωπαϊκές εταιρείε και επιχειρήσεις. Και αντλήσαμε και κάποια διδάγματα από την νομοθεσία αυτή. Καταρχήν, την περιμέναμε πώς και πώς και ήταν πολύ χρονοβόρεια διαδικασία. Κάναμε, μας πήρε πολύ καιρό να την ολοκληρώσαμε. Ήταν αρκετά επίμαχη και για μερικούς ε, ήταν σαν να επιβάλλονται υποχρεώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι προωθεί τι περαιτέρω καινοτομίε. Χρειάστηκε μία δεκαετία όμως για να καταλήξουμε στο αίσιο αποτέλεσμα του κανονισμού. Και μην ξεχνάμε ότι η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη βρίσκονται στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Σχεδίου και καλό είναι να επιταχύνουμε τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, ένα άλλο διδαγμα είναι ότι θα πρέπει όταν έχουν μειωθεί, καταργηθεί κάποια τέλη, να μην ε, αντικαθιστούνται από άλλου είδου τέλη, είτε είναι βασικά τέλη, είτε τίποτα άλλο. Να μην βγάζουμε από τη μία πλευρά και να βάζουμε από την άλλη δηλαδή. Επίσης, πότε αναμένεται αναθεώρηση, επανεξέταση του κανονισμού. Έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Γιατί το ΕΛΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό μια τέτοια αναθεώρηση του κανονισμού. Επίσης, για τις μελλοντικές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μπορούσαμε στις διαπραγματεύσεις να μεριμνήσουμε ώστε οι πολίτες μας να απολαμβάνουν περιαγωγή και εκεί χωρίς ε, επιπλέον χρεώσεις, με χρεώσεις εσωτερικού λοιπόν όπως είχε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Συλλεστών Δημοκρατών, η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι αυτή η έκθεση που μας παρουσιάζεται σχετικά με την λειτουργία της διάταξης για την κατάργηση της παραγωγής μας χαροποιεί πάρα πολύ. Γιατί είχαν μεγιστοποιηθεί, είχαν υπερτονιστεί πάρα πολύ κίνδυνοι και αν τα είχαμε λάβει όλα αυτά υπόψη μας, τελικά υποτίθεται θα αυξανόταν πολύ το κόστος, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ε, πολύ ε, βέβαια είχαν προβλέψει όλα αυτά για να ωφεληθούν ε, γιατί θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση. Και όπως είπε και η συνάδελφος, οι πολίτες είναι οι πρώτοι οι οποίοι έχουν επωφεληθεί. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς η εισαγωγή αυτής της διάταξη που δεν ήταν εύκολο. Εγώ ήμουν σκιώδη συγγήτρια, η συνάδελφος Πιλάρντε Καστήλιο ήταν η και θέλω να πω ότι μόνο με την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντάξει και της Επιτροπής για να είμαστε ειλικρινείς, το Συμβούλιο τελικά πέρα από τον Ιούλιο του 2017 ε, αποφάσισε να έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις και να αρχίσει να ισχύει η περιαγωγή. Αυτή ήταν λοιπόν μια κίνηση από τους Ευρωπαίους πολίτες και είχε και αποτέλεσμα οικονομικό. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που είναι πολύ περισμένες οι ρήτρε και για πρακτικές αθέμητες ε, και για ε, κάποια ε, καταφυγή σε θέματα ασφάλειας. Το θέμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανείς να μπορεί να ελέγχει κατά πόσον αυτό είναι νόμιμο ή όχι. Ως εκ τούτου, αυτό που έχει σημασία είναι ο Μπέρεκ ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, τοποθετηθούν σε αυτό το θέμα γιατί ο κανόνας θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά. Και επίσης ε, η αναθεώρηση θα πρέπει να προβλέψει και να εφαρμόσει έναν κανονισμό μόνιμης περιεγωγής. Εγώ θέλω να σας πω ότι θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Και νομίζω ίσως μπορούμε και να δώσουμε και μια πιο τυπική μορφή όταν τηλεφωνούμε εκ εκτός ε, της χώρας μας λέμε ότι ε, είναι σαν να τηλεφωνούμε ε, από το σπίτι μας. Αλλά τότε γιατί υπάρχουν αυτές, αυτό το επίθετο, ας πούμε, διεθνής κλίση. όταν μιλάμε για διεθνή κλίση, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το επίθετο, να λέμε ότι είναι στην Ευρώπη αυτές οι κλίσεις. Είναι λοιπόν μια ρύθμιση που θεωρώ ότι θα πρέπει και στις διεθνείς κλίσεις να ακολουθήσουμε τον δύο δρόμο όπως και στην περιαγωγή μέχρι να φτάσουμε στην κατάργηση. Άρα δηλαδή η δουλειά που έχετε αρχίσει να κάνετε για την εξέλιξη του κανονισμού ίσως την ίδια δουλειά θα πρέπει να αρχίσετε να κάνετε και για την κατάργηση των διεθνών κλήσεων. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα συμπληρωθεί πλήρως αυτός ο νέος κανονισμός. Έχουμε κάποιον από την ομάδα Renew Europe ε, για να αντικαταστήσει το συντονιστή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότητα τον κύριο Βέσα Τέραβα και να τον συγχαρώ και τον ίδιο και όσους ενεπλάξαν σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινήσαμε με την πρόταση 5-5-5, δηλαδή 5 λεπτά φωνητική για 5 μέρες το χρόνο και 5 μηνύματα SMS και 5 MB. Όχι δωρεάν, αλλά με, με χρέωση εσωτερικού, περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού. Και ξεκινήσαμε πολύ σοβαρές συζητήσει και είπαμε πλάκα μας κάνετε. Δράση είναι αυτή. Δεν είναι τίποτα. Και τελικά χαίρομαι γιατί καταφέραμε και καταλήξαμε σε συμφωνία. Όταν όμως ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια με τις, στις διαπραγματεύσεις, πολλοί φορεί εκμετάλλευση και πάροχοι υπηρεσιών είπαν ότι θα έπρεπε να αυξήσουν τις τιμές λιανικής σε εκείνους που δεν θα ταξιδέψουν ποτέ σε άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είπαν ότι πολλοί φορείς εκμετάλλευσης ε, δικτύου θα χρεοκοπήσουν και όπως ξέρουμε το 8% των Ευρωπαίων πολιτών μόνο ε, ε σε παρεκκλήσεις που ζήτησαν ε, και τώρα υπάρχει ένα όριο 14 κιλομπάιτ το μήνα. Αυτά είναι τα όρια που έχουμε επιβάλει μερικοί. Ερωτώ λοιπόν, έχουμε κάποιες πληροφορίες για κράτη-μέλη που πραγματικά χρειάστηκε να αυξηθεί την λενικής, η χρέωση λενικής για πολίτες που δεν κάνουν ποτέ ταξίδια σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πληροφορίες για φορείς εκμετάλλευσης ε, κινητών δικτύων που χρεοκόπησαν λόγω της ε, περιαγωγής με χρέος εσωτερικού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριος Μπόρκια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την παρουσίαση αυτή που ήταν πολύ συγκεκριμένη και πολύ επίκαιρη. Όντως, ε, ο κανονισμός αυτός ε, γνώρισε επιτυχία, σαφώς υπάρχουν θετικές επιπτώσεις και για τους χρήστες και για τις επιχειρήσεις. Και είναι πολύ θετικός ο κανονισμός για τη γενικότερη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό ότι μειώθηκαν οι τιμές και αυξήθηκε η κυκλοφορία των δεδομένων. Παρ' όλα αυτά όμως καθότι κινούνται θετικά τα πράγματα, μήπως θα πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα στις πτυχές εκείνες οι οποίες ε, θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω, προκειμένου ο κανονισμός αυτός να είναι ακόμα πιο θετικός, ακόμα πιο επικοδομητικός. Θα ήθελα να καταλάβω αν ε, οι φορείς εκμετάλλευσης αντέδρασαν τελικά θετικά σε όλα τα κράτη-μέλη ή αν είχαμε τελικά και κάποια ανομοιογένεια στις αντιδράσεις αυτές. Δηλαδή, κάποιοι φορείς εκμετάλλευσης σε ένα κράτος μέλος, ιδιαίτερα τουριστικό για παράδειγμα, βρέθηκε κάπως ζημιωμένος, καθότι υπήρχαν πάρα πολλοί τουρίστες που έκαναν χαρίσει περιαγωγή στο κράτος αυτό. Μία άλλη ερώτηση τώρα. Το 2015 είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης που είχαν αρχίσει να κοστολογούν συγκεκριμένε υπηρεσίες που κανονικά θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν και το κάνανε αυτό για να καταφέρουν τελικά να αντισταθμίσουν τα μειωμένα έσοδα που είχαν λόγω της περιεγωγής με χρέους εσωτερικού. Παρακολούθησε τα φαινόμενα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, υπήρχαν ορισμένοι καταναλωτές οι οποίοι δήλωσαν ότι πληρώσαν πολύ σημαντικές χρεώσεις. 30 Ιουνίου μας είπατε ότι θα εκπνεύσει ο κανονισμός αυτός. Επομένως, τι θα προκύψει από την δημόσια διαβούλευση. Μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν κάποιες αναδυόμενες, αν θέλετε, τάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδυόμενες απόψεις ή προσεγγίσεις αυτή τη στιγμή. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα και εγώ, να γνωρίζω αν από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποια είδη τοποθέτηση διαπραγματευτική απέναντι στον Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο και αυτό δεσμεύεται από τον καονισμό αυτό μέχρι το τέλο του, μέχρι να εκπνεύσει ουσιαστικά. Ποια είναι η στάση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει του Ευρωπαίου πολίτε. Και τώρα περάμε στους πράσινους. Υπάρχει κάποιος συντονιστής ή αναπληρωτής από τους πράσινους. Εγώ θα είμαι πιο συνοπτικός. Έχω δύο ερωτήσεις. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει πρόθεση ε, αναθεώρηση του κανονισμού, υποβολή νέου κανονισμού για την περιαγωγή. Ο νέος κανονισμός θα τροποποιήσει τον προηγούμενο ε, ή θα είναι τελείως καινούριο. Και μια και δεν έχουμε διαπιστώσει σημαντικό αντίκτυπο στους φορείς εκμετάλλευσης. Τι γίνεται με το όριο των, της, των τελών χονδρικής. Μήπως μπορούμε να μειώσουμε το το όριο, μια και δεν ε, υπάρχει αντίκτυπος. Ο κύριος Στοσενόφσκι. Σας ευχαριστώ. Ήμουν από τους σκιώδεις ηγητές που αναζητούσαν τρόπο για να είναι ο κανονισμός σύντομος, αποτελεσματικός και υγιής. Και χαίρομαι που βρήκαμε τελικά τη σωστή λύση έστω και μετά από πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι για τον κανονισμό γιατί είναι πολύ άρτιος και αυτό ισχύει και για τα όρια που τέθηκαν. Και χαίρομαι και για την επιτυχία που συνάντησε ο κανονισμός και στην εφαρμογή του. Και το λέω γιατί στην αρχή είχα αρκετούς εδιασμούς για τον κανονισμό. Πίστευα ότι θα υπάρξουν προβλήματα, θεωρούσα ότι θα δημιουργούσε δυσκολίες η εφαρμογή του, αλλά ευτυχώς τεύθηκε με επιτυχία. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, το 2022 θα λήξει η ισχύ του κανονισμού. Σίγουρα θα προηγηθούν σημαντικές δημόσιες και πολιτικές συζητήσεις και εδώ και αλλού. Και ο Μπερέκο, ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο και δυνατότητα να μειώσουμε ε, τη χρέωση χονδρικής. Μέχρι το 2022 μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Θα έχουμε τις τεχνολογίες πέμπτης γενιάς και πολύ σημαντικές επενδύσεις που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εκ των πραγμάτων, γιατί θα είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Οπότε, πώς προετοιμάζεστε για τη νέα κατάσταση. Θα έχουμε τεράστια αύξηση του όγκου δεδομένων και των παραμέτρων της περιαγωγής. Ξέρω ότι είναι κάπως πρόωρη ερώτηση, αλλά ποιες πιστεύετε θα είναι οι συνέπειες της νέας κατάστασης και πώς ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την περίοδο μετά το 2022, μετά την εκπνοή του κανονισμού. Πώς θα πλαισιώσει καλά αυτές τις νέες επενδύσεις. Δεν βλέπω κανέναν συντονιστή από την ΚΟΕ. Οπότε περνάμε στην υπόλοιπη ομιγύρια. Ο κύριος Κονσάλες Σέζαρες, όχι. Άλλος κανείς. Άλλος κανείς θέλει να λάβει μέρος στη συζήτηση. Όχι. Οπότε παρακαλώ τον κύριο Βέσα Τέροβα να απαντήσει και να καταλήξει και σε κάποια συμπεράσματα. Uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για τα σχόλια και χαίρομαι που όλοι συμφωνούμε ότι ο κανονισμός στέφθηκε με επιτυχία και συμφωνούμε σε πολλά επιμέρους σημεία. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον. Με ρωτήσατε τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την εκπνοή του κανονισμού τον Ιούνιο του 2022 και τι θα συμβεί με τη χρέωση χοντρικής, με τα τέλη χοντρικής και πώς θα λάβουμε υπόψη τεχνολογία 5G, τη μεγάλη αύξηση του όγκου των δεδομένων και τις ε, νέες επενδύσεις που θα χρειαστούν. Όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, βάσει των στοιχείων και των δεδομένων που έχουμε και των πληροφοριών από την έκθεσή μας και των στοιχείων που μας έχει δώσει ο Μπερέκ και τα κρατημέλη, τώρα αρχίζουμε και εκπονούμε μια μελέτη αντικτύπου και θα έχουμε και δημόσιες διαβουλεύσεις για να δούμε πώς θα προετοιμαστούμε για το μέλλον. Πάντως, το συμπέρασμα είναι ότι τίποτα δεν έχει αλλοιώσει την ανταγωνιστικότητα. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ότι η ανταγωνιστικότητα δεν έχει φύγει. Και μέχρι το τέλη του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει τα επόμενα της βήματα. Και αν το συμπέρασμα που θα καταλήξουμε θα είναι ότι θα χρειαστεί και περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση, δεν θέλω να το προεξοφλήσω αυτό το συμπέρασμα, θα υποβάλουμε την κατάλληλη πρόταση και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν επαρκή χρόνο να την εξετάσουν και ενδεχομένως να καταλήξουν σε συμφωνία. Επίσης, με ρωτήσατε πότε πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει για τα νέα ενδεχομένω ανατατόρια των τελών χονδρικής. Θα δούμε, θα εξαρτηθεί το χρονοδιάγραμμα της πρότασης από τις διαπραγματεύσεις ε, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Έχοντας υπόψη και το, την προθεσμία του Ιουνίου του 2022, που είναι η απότερη χρονική στιγμή ε, της απόφασης, αν αποφασιστεί τελικά, δηλαδή ότι θα χρειαστεί συνέχιση του κανονισμού ή ε, αναθεώρηση του κανονισμού στο μέλλον. Τώρα για τις τεχνολογίες πέμπτης γενιάς και τις επενδύσεις. Σίγουρα η περιαγωγή δεν είναι ένα μεμονωμένο θέμα, ξεχωριστό και απομονωμένο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλα ζητήματα. Ξέρω ότι πριν την περιαγωγή συζητήσατε θέματα της ασφάλειας για, το 5G. Επίσης, κατανομή του φάσματος ε, για τις τεχνολογίες πέμπτης γενιάς, σημαντικό θέμα. Και θα πρέπει να καταχωρηθεί το φάσμα στα 700 για το 26 μέχρι τα τέλη του έτους. Οπότε θα πρέπει να γίνουν και πολλές σημαντικές επενδύσεις στο μέλλον για να αναπτυχθούν μόνο ασφαλή δίκτυα 5G. Μόνο αυτά να παρουσιαστούν και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και κατά τη συζήτηση της περιαγωγής. Τώρα, για την ε, παράταση του κανονισμού της περιαγωγής και τι θα γίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο στις διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κανονισμός για την περιαγωγή είναι από τα εργαλεία της εσωτερικής αγοράς. Οπότε αν κανείς εντός της εσωτερικής αγοράς, επωφελείται από την απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Δηλαδή να μην υπάρχει πλέον χρέωση για την περιαγωγή. Τώρα, τι θα γίνει με τις τρίτες χώρες δεν αφορά τον κανονισμό της περιαγωγής. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις και για τα θέματα αυτά. Η κυρία Τόγια και ο κύριος Άνσιπ. Τι γίνεται με τις διεθνείς κλήσεις. Ξέρουμε ότι μετά τη συζήτηση, τη συζήτηση για το κώδικα της τηλεπικοινωνίας και τον κανονισμό για τον ΠΕΡΕΚ, και είναι όλο περίεργο, αλλά είναι στον κανονισμό του Μπερέκ. Εκεί αναφέρονται τα ε, ανώτατα όρια τιμολενικής για τι διεθνεί κλήσει. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει και υπάρχει και ρήτρα λήξη ισχύω. Και όταν οι νομοθέτε αποφασίσουν να επιλέξουν αυτό το θέμα, φυσικά διαφέρει από την αγορά της περιαγωγής, γιατί άλλο να κάνει κανείς κλήσεις στην χώρα και άλλος να κάνει διεθνή κλήση. Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες ε, υπηρεσίες επικοινωνιών μέσω του διαδικτύου που μπορεί να κάνει δωρεάν κλήσεις. Και γι' αυτό ακριβώς οι νομοθέτες αποφάσισαν να θεσπίσουν λιγότερο αυστηρούς κανόνες ε, για τις διεθνείς κλήσεις. Και για την ερώτηση του κυρίου Άσιπ, Έχουμε κάποια παραδείγματα. Με ρωτήσατε αύξηση των εγχώριων τιμών, των εθνικών τιμών. Πάντω, όπω σα είπα και στην παρουσίαση, η γενική παρατήρηση είναι ότι ακόμη και χώρε τιμέ ε, ακολουθούν φθήνουσα πορεία. Δεν ξέρω κάθε πάροχο ε, υπηρεσία κάθε φορέ εκμετάλλευση τι χρεώνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Πάντω, η γενική τάση είναι ότι ακόμη και χώρε τιμέ μειώνονται, μειώθηκαν. Οπότε η περιαγωγή και η περιαγωγή με χρέο εσωτερικού δεν επηρέασε τις εσωτερικές εγχώριε τιμέ. Επίσης, ε, μας ερωτήσετε κατά πόσο υπάρχουν παραδείγματα από περιπτώσεις όπου δεν προσφέρεται η περιαγωγή. Βεβαίως ε, και έχουμε παραδείγματα. Η περιαγωγή είναι μια εμπορική επιλογή του παρόχου, αλλά επειδή, όπως βλέπουμε από τα στατιστικά δεδομένα, ε, αρέσει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την περιαγωγή όταν ταξιδεύουν, προφανώς δεν είναι ενδιαφέρουσα η προσφορά αν δεν υπάρχει περιαγωγή. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα από ε, φορείς εκμετάλλευση δικτύου των κινητών επικοινών, τα MVNOs. Ε, αυτά όμως ε, είναι κάποια μεμονωμένα παραδείγματα. Δεν θα πρέπει να γενικεύουμε, γιατί δεν είναι μια ανταγωνιστική αυτή η προσφορά. Ο κύριος Πόκια ρώτησε ποια είναι η γενικά αντίδραση των παρόχων, ε, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών χοντρικής. Όπως είπα και στην αρχή, οι πάροχοι συμμορφώθηκαν με τους ε, κανόνες, με αυτά που αποφάσισαν οι νομοθέτες. Αποφάσισαν λοιπόν να ε, συμμορφωθούν. Αυτό εντάσσεται στον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό και βεβαίως ε, δέχτηκαν αυτή την ε, πολιτική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου ε, δεν ακούμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες από τους παρόχους, τουλάχιστον όχι περισσότερες από ό,τι ακούγαμε μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Βεβαίως οι επιπτώσεις στους παρόχους εξαρτώνται από το κατά πόσον κανείς είναι καθαρός αποδέκτης ή καθαρός αποστολέας των ε, ε, δεδομένων της επικοινωνία. Στους ανθρώπους αρέσει να ταξιδεύουν σε καλύτερες συνθήκες και ακόμα και στις χώρες εκείνες όπου εξετάζει κανείς συγκεκριμένα δεδομένα για ε, τιμές ε, χονδρικής και αν συγκρίνει κανείς ε, αυτές τις τιμές, αυτά τα τέλη με ρυθμιζόμενα τέλη, είναι πιο κάτω, που σημαίνει ότι οι πάροχοι μπορούν να καλύψουν ε, το κόστος της χοντρικής Και αν δει κανείς και τις χώρες όπου τουλάχιστον ακόμα δεν έχει διαδοθεί η περιεγωγή. Εκεί όπου οι πάροχοι πληρώνουν ε, υψηλά τέλη περιεγωγής. Αν δει κανείς τις εταιρείες ε, που έχουν ζητήσει, έχουν αιτηθεί την παρέκκληση βιωσιμότητας ή ε, χρησιμοποιούν πιο συχνά την εύλογη χρήση. Θα διαπιστώσει κανείς ότι σε αυτές τις χώρες βλέπουμε να εφαρμόζεται η παρέκκληση βιωσιμότητας. Βλέπουμε όμως μια τάση όπου όλο και λιγότεροι ε, πάροχοι βασίζονται ή καταφεύγουν στην ε, βιωσιμότητα. Οι πάροχοι καταλήγουν σε συμφωνίες που, τις τους επιτρέπουν να προσφέρουν υπηρεσίες λιανικής χωρίς ε, να ε, ζημιώνονται ουσιαστικά. Υπάρχουν βέβαια ε, διαφορές στις διάφορες χώρες, αλλά αυτή είναι η γενική εικόνα. Βεβαίως το τι θα συμβεί στο μέλλον, αυτό θα φανεί. Νομίζω ότι κάλυψα τις ερωτήσεις και αυτά είχα να σας πω. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς ε, να διατυπώσει κάποια άλλη ερώτηση. Αν όχι, ε, έκλεισε και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που είναι μεγάλη επιτυχία για μας. Γιατί ακόμα και πολίτες ε, που δεν ε, ε, είναι ενθουσιασμένοι ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η περιεγωγή είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για τη σημερινή συνεδρίαση. Ενημέρωση από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 14η Σύνοδο του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Πρόκειται για μια αποστολή του αντιπροσωπείου που συμμετείχαν συνάδελφοι από διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές πέρα από την δική μας επιτροπή. Είχαμε και εκπροσώπηση από την ΙΜΚΟ, Γιούρι, Λίμπε, Κούλτερ αλλά και από τη ΣΤΟΑ. Και έλαβε χώρα η συνεδρίαση αυτή από τις 25-29 Νοεμβρίου του 2019. Η διάσκεψη των Προέδρων είχε δώσει το δικαίωμα σε 10 μέλη να ενταχθούν στην αποστολή αυτή, αλλά εν τέλει, επειδή το φόρουμ αυτό συνεδρίασε παράλληλα με την Ολομέλεια του Στρασβούργου τον Νοέμβριο, είχαμε τελικά τέσσερα μόνο μέλη, τέσσερις ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στο φόρουμ αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από την επικεφαλής αντιπροσωπείας, την κυρία Γκάλβες Μούνιος, να μας ενημερώσει εν συντομία για την αντιπροσωπεία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Φόρουμ για την Κυβέρνηση Διαδικτύου είναι ένα φόρουμ για ένα διάλογο όσον αφορά την δημόσια διακυβέρνηση του διαδικτύου. Η 14η αυτή συνεδρίαση έλαβε χώρα στο Βερολίνο από τις 25-29 Νοεμβρίου του 2019 και το βασικό θέμα ήταν ένας κόσμος, ένα διαδίκτυο, ένα κοινό όραμα. Τα βασικά θέματα την διακυβέρνηση των δεδομένων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η ανθεκτικότητα σε επιθέσεις, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαρτιζόταν προφανώς από την υπομφαινόμενη, από την Μαρίνα Καλιουράντ, από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, από την Κάρεν Μέλχιορ, από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και από την Αλεξάνδρα Γκίζε, από την Επιτροπή Εσωτερικών, Εσωτερικής Αγοράς. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, διοργανώθηκε το φόρουμ αυτό παράλληλα με την Ολομέλεια του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα τελικά να μην έχουμε την ευκταία συμμετοχή και έπρεπε επίσης πολλοί συνάδελφοι να ψηφίσουν για μια σημαντική πρόταση στα πλαίσια της Ολομέλειας του Νοεμβρίου. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε στο πλαίσιο του φόρουμ αυτό να αυξήσουμε την κοινοβουλευτική πτυχή και να καλέσουμε όλο και περισσότερους βουλευτές, καθώς επίσης και εκπροσώπους του Global South. Το φόρουμ αυτό διοργανώθηκε από την Αιγίδα των ΗΕ και Γενικό Γραμματέα των Εθνών, πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στο στις αναδυόμενες αυτές τάσεις αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτών μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ε, εκμετάλλευση αθέμητη και παράνομη πολλών δεδομένων η οποία στρέφει τους πολίτες ε, τους μεν αντίον των δε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε έναν απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών, πράγμα το οποίο θα λάβει η χώρα, προκειμένου να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ένα διεθνές πλαίσιο. Η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ είπε ότι η πολυμέρεια αποτελεί πραγματικά τη βασική αρχή για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Τόνισε επίσης ακόμα ότι όλοι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον πυρήνα του διαδικτύου ως κοινό καλό, κοινό αγαθό, καθότι επηρεάζει θετικά τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα. Δεν μπορεί λοιπόν να διαμορφώνεται το διαδίκτυο μόνο από τις κυβερνήσεις και τα κράτη. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχε στην πολύ ζωντανή συζήτηση που έγινε με άλλους βουλευτές από όλο τον κόσμο, όπου συζητήσαμε πρώτον την τεχνητή νοημοσύνη, δεύτερον τη διεθνή συνεργασία για ένα πιο ανοιχτό, πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο διαδίκτυο και τρίτον το ζήτημα των δημοκρατιών στην ψηφιακή εποχή και το ρόλο των κοινωνικών δικτύων, των δικτύων κοινωνικής ε, δικτύωσης. Επίσης, αναφερθήκαμε και στις κρίσιμες υποδομές. Επίσης, ε, συναντήσαμε και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως μία από την Νότια Αφρική, που ενθαρρύνει νέα κορίτσια να μαθαίνουν νέες γλώσσες πληροφορικής και τον κώδικα πληροφορικής. Επίσης, Υπόθηκε στα πλαίσια του φόρουμ αυτού ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί διακριτική μεταχείριση. Πολύ συχνά και στον τομέα αυτό της πληροφορικής και της τεχνικής νοημοσύνης υπάρχει ε, διακριτική μεταχείριση κατά των ε, μαύρων. Επίσης, υπόθηκε ότι θα πρέπει, να καταπολεμηθεί κάθε διακριτική μεταχείριση που έχει να βάση του φύλου όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση στον κώδικα. Ήδη από το 2005 ο λεγόμενος ε, πατέρας της πληροφορικής ασχολείται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριο Σέρφ μα είπε ότι ο όρο τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη από τη δεκαετία του 60, αλλά ότι ακόμα απέχουμε πάρα πολύ από το να έχουμε μια πραγματική τεχνητή νοημοσύνη. Αποσαφήνισε ότι απαιτείται ακόμα να γίνει πολλή έρευνα και ως παράδειγμα τόνισε την αυτόματη μετάφραση, η οποία δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την τεχνητή αυτή αυτόματη μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη. Όπως σας είπε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και θα πρέπει να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της τεχνητής νομοσύνης ακόμα και κοινωνιολόγοι. Επίσης, Συζητήσαμε με την ICON, με την αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με το κίνημα νεότητος ΑΕΖΕ. Και ολοκληρώνοντα την παρουσίασή μου αυτή, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέκρινε την, το κλείσιμο του διαδικτύου και την απαγόρευση χρησιμοποίησης ε, του διαδικτύου από ορισμένου πολίτες ή τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως μέσο καταστολής. Είπε επίση ότι θα πρέπει όλοι να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθότι το διαδίκτυο επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινή ζωή των πολιτών και επηρεάζει τελικά και την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατιών, αλλά και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και την επιτυχία των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Τρίτον, τονίσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ψηφιακές τεχνολογίες για να πετύχουμε τους στόχους τη βιωσιμότητα. Τέταρτον, τονίσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε πρότυπα υψή τη ποιότητα, όπως το GDPR, προκειμένου να καταφέρουμε να υπερβούμε τις δυσκολίες όσον αφορά τη θέσπιση διεθνών κανονισμών. Και τέλος, να ευχαριστήσω τον Χόλγκαν Γκβένσιν, ο οποίος ήταν, αν θέλετε, ο μέντοράς μας για την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να τον ευχαριστήσω όλος ιδιαιτέρως, γιατί ε, εγώ ήμουνα ακόμα τραυματισμένη όταν ήμουνα στο Βερολίνο και με βοήθησε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θέλει κανείς άλλο το λόγο για να σχολιάσει αυτή την αποστολή στο Βερολίνο. Όχι. Οπότε σας ευχαριστώ και να σας πω ότι το επόμενο φόρουμ ε, διακυβέρνησης του διαδικτύου θα λάβει χώρα στο Κατοβίτσε, στην Πολωνία, 2 με 6 Νοεμβρίου. Αυτά ευχαριστούμε για την ενημέρωση την κυρία Γκάλβες Μουνιός και ολοκληρώσαμε τις απογευματινές μας εργασίες. Γεια σας.